Allora, cominciamo Ας αρχίσουμε λοιπόν γιατί έχουμε καθυστερήσει. Για το σημείο 3 της ημερήσιας ε, διάταξης, της γλώσσας της γνωρίζετε, έγινε το web streaming. Ε, μου ανακοινώθηκε ότι υπάρχουν 10 μέλη της αντιπροσωπείας της ε, από το Κοινοβούλιο Μέρκο Σουρ ε, που επισκέπτονται το Κοινοβούλιο 21 με 23 Ιουνίου και είναι παρόντες στη συνεδρίασή μας, τους καλωσορίζω. Στο σημείο 4 της ημερήσιας διάταξης έχουμε την επίσκεψη της κοινή με την Επιτροπή ε, των Προϋπολογισμών Αντιπροσωπείας στην Κροατία, 22 με 25 Ιουνίου στην Κροατία θα γίνει η επισκέψη αυτή. Όσον αφορά την αντιπροσωπεία για την Κροατία, η Επιτροπή έδωσε στοιχεία που μπορεί να είναι χρήσιμα για τις αντιπροσωπείες. Είναι παρούσα η Επιτροπή. Ε, αν θέλετε να δώσετε κάποιες πληρωματικές πληροφορίες στην Επιτροπή μας, σας δίνω το λόγο. Διαφορετικά μπορούμε να προχωρήσουμε με την ημερήσια διάταξη. Τίποτα λοιπόν δεν έχετε να πείτε. Εντάξει λοιπόν, προχωρούμε επειδή έχουμε καθυστερήσει και έτσι κερδίζουμε λίγο χρόνο. Ας περάσουμε τώρα στα σημεία 8, 9 και 10 της ημερήσιας διάταξης. Αφορά ε, την Ευρωπαϊκή, αφορούν τα σημεία αυτά την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Λίγη ησυχία παρακαλώ. Ε, επ' αυτού, λίγο πριν από την ε, συνεδρίαση της Επιτροπής μας μου δόθηκε ένα σημείωμα εκ μέρους της ε, Γραμματείας που αναφέρεται στο γεγονός ότι ε, έχουν δοθεί ανεπίσημα τα σχετικά έγγραφα μετά την ε, πολιτική συμφωνία ανάμεσα στην Κομισιόν, το Συμβούλιο, την ε, είπα, εκπρόσωπο, κυρία Άστον, ε, και τη συνεδρίαση που έγινε στη Μαδρίτη, φαίνεται ότι η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων ΑΦΕΤ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, μπόρεσε να εγκρίνει τη σχετική ε, θα μπορέσει να ε, ε, εγκρίνει τη σχετική έκθεση στη συνεδρίασή της στις 14 Ιουλίου. Έτσι όλες οι επιτροπές που θα πρέπει να γνωμοδοτήσουν θα πρέπει να είναι έτοιμες να υιοθετήσουν τις γνωμοδοτήσεις τους πριν από τις 14 Ιουλίου. Κατά συνέπεια λοιπόν η Επιτροπή μας, η ΚΟΝΤ, θα πρέπει να υιοθετήσει την ε, γνωμοδότησή της στην τελευταία της συνεδρίαση πριν από το καλοκαίρι που όπως ξέρετε θα γίνει στις 12 Ιουλίου. Αυτό σημαίνει, αν λάβουμε υπόψη μας και τις μεταφράσεις κλπ, ότι η τελική προθεσμία για την υποβολή ε, ε, τροπολογιών ε, είναι μέχρι την Πέμπτη στις 12 η ώρα αυτή την εβδομάδα. Διαφορετικά δεν θα μπορέσουμε να συμβάλλουμε και να έχουμε συμμετοχή στις εργασίες που διεξάγει η Επιτροπή ΑΦΕΤ. Αυτά λοιπόν για τα σημεία 8, 9 και 10 της σημερινής διάταξης. Για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης δίνω τώρα το λόγο στον ε, κύριο Κάλφιν, τον εισηγητή. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Δεν θα μακρηγορήσω, διότι την τελευταία φορά θα θυμούνται ίσως οι συνάδελφοι ότι ουσιαστικά παρουσίασα ένα κείμενο χωρίς να το έχω όμως παρουσιάσει υπόψη, να το θέσω επισήμως υπόψη των μελών, γιατί είχαμε αποφασίσει να μην ξεκινήσουμε κάποια διαδικασία προτού έχουμε τις ε, σχετικές προτάσεις της Κομισιόν για την ΕΙΕΔ. Αυτό λοιπόν είναι το πλαίσιο, η έκθεση πλαίσιο για τη σύσταση της ΕΕ της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, με καθήλυνα αρμόδια την Επιτροπή ΑΦΕΤ, η ε, κύριοι ε, Μπρόκ και Φερχόφστατ ε, και είναι οι συνήθεις ηγητές, ο κύριος Φερχόφστατ είναι ΑΦΚΟ. Και πριν την καλοκαιρινή διακοπή θα πρέπει να έχει συζητηθεί στο Κοινοβούλιο. Ξέρουμε ότι πλέον το Κοινοβούλιο έχει την εξουσία της συναπόφασης Έχουμε τον τροποποιητικό κανονισμό, τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης και τον δημοσιονομικό κανονισμό σε σχέση με αυτή την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία. Σε ό,τι αφορά την έκθεση Brock Brockfer-Hofstadt... έχοντας πλέον όλα τα έγγραφα στη διάθεσή μας και έχοντας ε, κάνει στον ε, τετραμερή διάλογο πολύ εντατικέ συζητήσεις, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Συμβούλιο, Κοινοβούλιο και το γραφείο της ε, είπα της εκπροσώπου έχουμε μια σαφή ιδέα για το τι γίνεται και το τι δεν γίνεται. Μέχρι χθε, συγκεκριμένα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επέμενε ο προϋπολογισμός της ΕΙΕΔ να σχετίζεται, να συνδέεται με τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ώστε να χρησιμοποιούνται ήδη γνωστές διαδικασίες και για την έγκριση και για τον έλεγχο του προπολογισμού φαίνεται ότι αυτό δεν είναι δυνατόν. Υπήρξε κάθετη αντίδραση και διαφωνία από το Συμβούλιο. Επομένως τώρα, από ό,τι φαίνεται, θα υπάρχει ξεχωριστός προϋπολογισμός για την ΕΕΔ υποξεχωριστό τίτλο, παρθμόν 6. Αυτός ο προϋπολογισμός θα αφορά μόνο τις διοικητικές δαπάνες της ΕΕΔ ενώ οι επιχειρησιακές δαπάνες ε, θα βαρύνουν την Κομισιόν. Επομένως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έχει πλήρες δικαίωμα απαλλαγής για τον προϋπολογισμό της ΕΕΔ. Όπως ισχύει για τους εκπαιδευτικούς οργανισμούς Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα γίνεται απαλλαγή και για τις διοικητικές δαπάνες. αυτό που ενδιαφέρει την Επιτροπή μας είναι ότι θα έχουμε την απαλλαγή για τις επιχειρησιακές δαπάνες στο πλαίσιο της διαδικασίας απαλλαγής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό θα δημιουργήσει κάποια προβλήματα σε ό,τι αφορά την Επιτροπή Προπολογισμού. Επομένως, επιμείναμε εντόνως και υπήρξε για Γενική Συμφωνία η, Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ένα έγγραφο στο οποίο θα εμφανίζονται όλες οι δαπάνες που σχετίζονται με την ΕΙΕΔ ή δυνατόν για τη διαδικασία έγκριση του προπολογισμού του επόμενου έτου, όταν δηλαδή έχει ξεκινήσει στο Κοινοβούλιο αυτή η διαδικασία. Έτσι το Κοινοβούλιο θα έχει μια γενική εικόνα για τι δαπάνε οι οποίε σχετίζονται με τι εξωτερικέ δράσει. Υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα, το οποίο είναι πολύ σημαντικό για μας. Συγκεκριμένα πρόκειται για την ευθύνη, για την αρμοδιότητα για την απαλλαγή. Επειδή υπάρχει μία μετάθεση, μετατόπιση εξουσίας μεταξύ κομισιών, ΕΙΕΔ, στις διάφορες φάσεις της διαδικασίας κατάρτισης του και έγκρισης του προπολογισμού, υπάρχει ο κίνδυνος να μην έχουμε σαφή ευθύνη σε ό,τι αφορά την απαλλαγή. Δηλαδή, σε ό,τι αφορά το σχεδιασμό των δαπανών που προέρχεται από την ΙΕΘ. Η υλοποίηση είναι αρμοδιότητα της Κομισιόν και αυτή δίνει εντολή στον επικεφαλής της ε, αντιπροσωπείας, ο οποίος ορίζεται από την ΙΕΔ για να υλοποιήσει τον προϋπολογισμό. Πώς καταλαβαίνετε αυτό δημιουργεί ε, αρκετές ε, θέσεις, υπάρχουν αρκετοί υπάλληλοι οι οποίοι εμπλέκονται και ίσως κάποιος ε, θεωρήσει ή υποκριθεί ότι δεν υπάρχει σαφής αρμοδιότητα και ευθύνη σε αυτή τη ε, μετάθεση αρμοδιοτήτων και ευθυνών μεταξύ διαφόρων ε, υπαλλήλων των θεσμικών οργάνων. Θα πρότεινα λοιπόν και φαντάζομαι ότι θα καλωσορίσει η υποκριθει οτι δεν υπαρχει σαφη αρμοδιοτητα και ευθυνη σε αυτη τη μεταθεση αρμοδιοτητων και ευθυνων μεταξυ διαφορων υπαλληλων των θεσμικων οργανων θα προτεινα λοιπον και φανταζομαι οτι θα καλωσορισει η κομισιον την προσέγγιση αυτή να δημιουργήσουμε ένα σύστημα διασφαλίσεων, ασφαλιστικών δικλείδων, ώστε να μην ακούσουμε την Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού την εξήγηση ότι κάποιο δεν μπορεί να είναι υπόλογο ή υπεύθυνο επειδή έχουν αλλάξει οι αρμοδιότητες. Και υπάρχουν κάποιες καλές ιδέες, οποίες θα μπορούσαμε να προτείνουμε, ώστε η Επιτροπή, η οποία θα είναι ε, η αρμόδια για τις επιχειρησιακές δαπάνες, να έχει τον πλήρη έλεγχο και την πλήρη βέβαια εμπιστοσύνη. Στο βαθμό που, που υλοποιείται ο προϋπολογισμός για τις συγκεκριμένες δαπάνες. Υπήρξε επίσης ένα θέμα σε σχέση με τον εσωτερικό έλεγχο στη συμφωνία, η οποία την οποία πετύχαμε χθε, υπήρξαν κάποια ζητήματα που σχετίζονται με την Όλαφ και δέσμευση Επιτροπής ε, της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης και των κρατών μελών να διευκολύνουν και να βοηθήσουν την Όλαφ στο έργο της. Υπήρξαν κάποια ζητήματα σε ό,τι αφορά το εσωτερικό έλεγχο, το internal audit. Για μένα δεν είναι πολύ ξεκάθαρα τα πράγματα. Εσωτερικό έλεγχο τη Επιτροπή και εσωτερικό ε, έλεγχο ε, τη ΕΙΕΔ. Θα υπάρχει συνεργασία μεταξύ των δύο φορέων για την έλεγχο των επιχειρησιακών δαπανών. Νομίζω ότι θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι ο εσωτερικό έλεγχο τη Επιτροπή, εφόσον αυτή είναι αρμόδια για τον επιχειρησιακό προπολογισμό, θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να προβαίνει σε κάθε είδου ελέγχους ε, και μελέτε και έρευνε. εντός ε, του πεδίου εφαρμογής ε, των επιχειρησιακών δαπανών επικεφαλής της αντιπροσωπείας. Τώρα, υπάρχει μια συγκεκριμένη διατύπωση που δεν ξέρω από πού ακριβώς ε, προήλθε. Ίσως θα ήταν καλό να έχουμε κάποια ανταλλαγή απόψεων. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα ορθού ελέγχου των κονδυλίων που δαπανώνται από την ΕΙΕΔ, έλεγχο από πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, υπάρχουν κάποια ζητήματα δεν νομίζω ότι είναι απαραίτητο να τα θέσουμε σήμερα. Είναι ελάσσον σημασίας. Παραδείγματο χάρη η ευθύνη των επικεφαλής αντιπροσωπιών ή των ε, προσωρινών ε, υπαλλήλων, των εκπροσώπων δηλαδή των κρατών μελών ε, στην υπηρεσία εφόσον και εγκαταλείψουν την υπηρεσία. Να πρέπει να είναι δηλαδή υπεύθυνοι για, τη δράση τους και τις πράξεις τους για όσο διάστημα ήταν στην υπηρεσία. Νομίζω ότι θα έχουμε κάποιες ε, σαφείς απαντήσεις και δεν χρειάζεται να επισέλθουμε τώρα σε λεπτομέρειες. Τέλος, σε ό,τι αφορά τη διαδικασία. Για να ξεκινήσει η διαδικασία όπως προτείνατε κύριε Πρόεδρε και για να έχουμε επισήμως τη δυνατότητα τροποποίησης, υποβολής ε, τροπολογιών, σας υποβάλλω το σχέδιο γνωμοδότησης που είχα παρουσιάσει στην προηγούμενη συνεδρίαση δεν είναι πλήρως ενημερωμένη, δηλαδή με βάση τις συνομιλίε που είχαμε μέχρι τώρα. Υπάρχει όμω όλε τι γλώσσε τουλάχιστον και άρα μπορούμε να ξεκινήσουμε τη διαδικασία κατάθεση τροπολογιών. Εγώ από πλευρά μου θα κάνω και εγώ κάποιε τροπολογίε. Κάποιε ε, ήδη αυτή τη στιγμή ε, διανέμονται ε, στα μέλη τη Επιτροπή. Και έτσι θα εμπλουτίσουμε και το σχέδιο της νομοδότησης και με τα αποτελέσματα του χθεσινών διαπραγματεύσεων του τραμερού διαλόγου. Νομίζω ότι αυτά είναι από την πλευρά της Επιτροπής μας. Νομίζω ότι μπορούμε να καταλήξουμε πριν την ΑΦΕΤ με τη δική μας γνωμοδότηση για να περιμένουμε την ψηφοφορία τον Ιούλιο. Σίγουρα θα έχουμε πολλή δουλειά όταν χρειαστεί να δούμε τα άλλα τμήματα της απόφασης και δει το δημοσιονομικό κανονισμό που το φθινόπωρο θα χρειαστεί στην Επιτροπή μας να τον μελετήσουμε. Ευχαριστώ. Εσλέ, ευχαριστώ πάρα πολύ να πω πως ο κύριος Κάλφιν θα πρέπει να επικαιροποιήσει την παλαιά πρόταση γιατί αυτό το οποίο έχουμε μπροστά μας είναι μια παλαιά πρόταση και έχει περάσει ο χρόνος και έχουμε όλες αυτές τις τροπολίες λογίες. Οπότε καλύτερο θα ήταν, γιατί είναι δύσκολο για όλους εμάς, εσείς να λάβετε υπόψη τις νέες τροπολογίες από χτες, γιατί αυτά τα οποία είναι τώρα μπροστά μας δεν μας βοηθούν. Θα καθόμαστε να ασχολούμαστε άδικα. Γι' αυτό σας παρακαλώ εσείς να α, τα αποσύρετε και να την επικαιροποιήσετε για να μην γίνει και η Επιτροπή μας καταγέλαστη. Δεν είναι δυνατόν να κινούμαστε έτσι. Υπό το φως των νέων ε, εξελίξεων. Οπότε νομίζω πως αυτά τα οποία έχουμε μπροστά μας πρέπει να αλλάξουν σε κάνα δύο σημεία ε, και κατά τα λοιπά μπορούν νομίζω να ε, υποβληθούν και να υποβληθούν στην Επιτροπή και να υποβληθούν και τροπολογίες. Σε όλες τις συνεδριάσεις οποίες έλαβα μέρος και αυτή είναι η τρίτη συνεδρίαση σήμερα όσον αφορά την ΑΕΔ. Παντού είπανε πως θα πρέπει να φεθεί στις ομάδες το αν θα ψηφιστεί η έκθεση Μπροκ ήδη τον Ιούλιο. Οπότε έχετε χρόνο να επεξεργαστείτε ξανά νομίζω την έκθεσή σας εδώ πέρα για να μην έχουμε και εμείς να κάνουμε με ένα πράγμα το οποίο δεν καλύπτει τα βασικά πράγματα του δημοσιονομικού ελέγχου. Κάντε μας λοιπόν αυτή τη χάρη και κάντε μόνοι σας, μόνος σας αυτή τη δουλειά. Έχουν διαπραγματευτεί ενω μεταξύ και άλλα πράγματα. Έχει αλλάξει η κατάσταση και θα οδηγήσει αυτό μόνο σε σύγχυση και χάος. Νομίζω και η γραμματεία μπορεί να σας βοηθήσει για να ε, είναι και καθαρά τα, τα πράγματα π.χ. στο σημείο 3-4 όπου πρέπει να επιμείνουμε πως ε, οι εσωτερικοί ελεκτές κομισιών προσεχώς θα πρέπει να είναι υπεύθυνοι και για την ΕΙΕΔ. Γιατί ξέρετε πως και με τις άλλες αποκεντρωμένες υπηρεσίες έχουμε πολύ καλές εμπειρίες ε, μέχρι στιγμής. Οπότε επειδή μας απασχολεί πάρα πολύ αυτό το, το πράγμα ως Επιτροπή Πολιτισμού, παρακαλώ να το δείτε. Ευχαριστώ. Grazie, onorevole Gaier. Gaier. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ένα ερώτημα προς εσάς. Μόλις είπατε πως πρέπει να λάβουμε την απόφαση στις 12 Ιουλίου. Είμαστε σε μια λίγο επισφαλή κατάσταση γιατί αφενός προετοιμαζόμαστε για μια διαδικασία για την οποία δεν ξέρουμε πότε θα εισαχθεί και από την άλλη έχουμε προθεσμίες. Οπότε η πρόκληση όπως την κατάλαβα εγώ είναι η εξής. Έχουμε ένα πιθανό νομικό πλαίσιο για την υπηρεσία ε, στο οποίο συνεννοήθηκαν χτες τα τέσσερα μέρη που διαπραγματεύονται και εκεί πέρα εξασφαλίζονται τα δικαιώματα μας τα κοινοβουλευτικά όσον αφορά την λήψη αποφάσεων και στην περίπτωση που θέλουμε να γίνει η αλλαγή του προϋπολογισμού και όσον αφορά τον κανονισμό του προσωπικού. Διαφυλάσσονται τα δικαιώματά μας. Αυτό σημαίνει πως θα πρέπει να προετοιμαστούμε έγκαιρα να εκφράσουμε την άποψή μα ω Επιτροπή Ελεγχτού Προεπλογισμού για την έκθεση Μπρόκα. Αν όμως με ενημερώνουν σωστά, τότε 12 Ιουλίου είναι πολύ αργά γιατί θα, είναι η... γιατί θα γίνει στην τελευταία Ολομέλεια του Ιουνίου. Εάν ισχύει κάτι τέτοιο, το θέμα είναι τι θα γίνει με την ε, διαδικασία. ο συνάδελφο ο κύριο Κάλφιν έχει επεξεργαστεί κάποια πράγματα. Είπαμε να μην τα δούμε μέχρι να είναι τα πράγματα ξεκάθαρα, οπότε να μην ε, κοιτάμε το φάκελο άσκοπα. Τώρα λοιπόν έχουμε ένα μικρό προβληματάκι. Το θέμα είναι αν εμείς με το έγγραφο της 11ης ε, Πέμπτου μήπως μπορούμε να κάνουμε μια ενοποιημένη έκδοση η οποία θα μας δώσει δυνατότητα μέχρι την Παρασκευή πράγματι να γράψουμε τροπολογίες. Αυτή είναι μια διαδικασία ε, που θα μπορούσε να την κάνει και ο Ιβάιλο Κάλφιν ο ίδιος για τα σημαντικά πράγματα αλλά και εμείς ως ε, συντονιστές που ε, είμαστε μαθημένοι σε αυτά τα πράγματα. Εάν θέλουμε λοιπόν μπορούμε να το κάνουμε κάπως γρήγορα, να συμφωνήσουμε και στην ανάγκη να καταθέσουμε κοινέ τροπολογίε. Το πρώτο ερώτημα είναι λοιπόν, έχω καταλάβει σωστά όσον αφορά την 12η ε, ότι ίσως είναι πολύ μακριά και δεν προλαβαίνουμε. Και το δεύτερο ερώτημα δίνεται σε όλους μας στην Επιτροπή. Εάν μπορεί να ενοποιηθεί το έγγραφο και μου φαίνεται ότι είναι ζήτημα copy-paste και όχι πολιτικής σκέψης. Μήπως λοιπόν τότε θα είναι δυνατόν να έχουμε μια ενοποιημένη έκδοση για να μπορέσουμε να συνεννοηθούμε μέχρι την Παρασκευή για τροπολογίες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Επαναλαμβάνω αυτό που σας είπα πριν. Μία ώρα πριν από την σημερινή μας συνεδρίαση έλαβα ένα σημείωμα από τη γραμματεία το οποίο μου έδινε την εξής πληροφορία ότι μέσω της συμφωνίας που επιτέχθη χθε στη Μαδρίτη η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ΑΦΕΤ, θα λάβει απόφαση για το θέμα αυτό που συζητάμε, δηλαδή για την ε, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση στι 14 Ιουλίου. Αυτό σημαίνει ότι οι γνωμοδοτήσει των ενδιαφερομένων ε, επιτροπών πρέπει να είναι διαθέσιμε νωρίτερα. Η γραμματεία λοιπόν με ενημερώνει ότι η δικιά μας γνωμοδότηση πρέπει να είναι έτοιμη μέχρι τις 12 Ιουλίου. Και η πρόταση που κάνει η γραμματεία για να μπορέσουμε να γνωμοδοτήσουμε στις 12 Ιουλίου, η τελική προθεσμία για τις ε, τροπολογίες είναι 25 Ιουνίου 12 η ώρα. Θα πρέπει λοιπόν σήμερα να πάρουμε μια απόφαση σχετικά με το πώς θα προχωρήσουμε, γιατί όντως είναι περιορισμένα τα χρονικά περιθώρια που έχουμε. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε πώς θα προχωρήσουμε σε σχέση με αυτές τις ε, ημερομηνίες και αυτές τις προθεσμίες που σήμερα τις ε, ε, μάθαμε κι εμείς. Υπευλήθη ένα σχέδιο και στην Επιτροπή Προπολογισμού, χωρίς προθεσμία τροπολογιών. Ε, είναι χάλια η διαδικασία. Εμείς τι κάνουμε εδώ πέρα. Δεν θέλω εγώ να λάβω μέρο. Εντάξει να πάμε γρήγορα, αλλά δεν ανάγκη να τσακιστούμε και να αρχίσουμε να κάνουμε copy-paste κτλ. Είναι 32 σελίδες. Εγώ θέλω να επεξεργαστώ πλήρως την ε, πρόταση ε, ευθύς εξ αρχής. Εκεί πέρα στα σημεία στα οποία αφορά την απαλλαγή και τον έλεγχο του προπολογισμού πρέπει να τα ξαναδούμε. Γι' αυτό σας παρακαλώ ο κύριος ε, Κάλφιν ε, να κάνει μια πρόταση στα αγγλικά, επικαιροποιημένη για να μπορέσουμε. Δεν χρειάζονται καν τροπολογίες. Θέλω να σου πω εγώ τι θέλω να διαγραφεί και για μένα έχει λήξει το, το ζήτημα. θα χρειαστεί να, να κάνουμε 30 τροπολογίες. Γιατί να το κάνουμε έτσι τόσο είναι και μια συμφωνία που δεν μας δεσμεύει. Ούτως ή άλλως έχουμε πει πως θέλουμε να, αποφύγει, να αποφύγουμε αυτή τη διαδικασία, να έχουμε μια τακτική και κανονική διαδικασία λήψη αποφάσεων. Να, να δούμε και ποιος θα είναι αυτός ο διοικητικός ε, προϋπολογισμός. γιατί μιλάμε για 10 εκατομμύρια ευρώ επιχειρηματικό, επιχειρησιακό, ήταν 10 εκατομμύρια ευρώ για τι τις θέσει, αλλά συνολικά ο διοικητικό προπολογισμό πώ θα κοστίσουν μετά αυτές τις θέσεις. Δεν το ξέρει κανείς. Θα ήθελα λοιπόν, εάν έχετε την ε, βάση διαβούλευση του συναδέλφου Γκαλτιέρη, δεν νομίζω, μπορούμε να σβήσουμε 3-4 σημεία για να φύγουν, να έρθουν και οι παρεξηγήσεις και να συνεχίσουμε ούτως ή άλλως ε, το ζήτημα αυτό θα ε, συζητηθεί πιο ουσιαστικά στην Επιτροπή Προπολογισμού. Για να μην κάνουμε και δουλειά τζάμπα. Και δεν υπάρχει και καμία ούτως ή άλλως προθεσμία γιατί περιμένουμε τις ομάδες να δούμε τι θα γίνει με την έκθεση Μπροκ και στην ανάγκη θα γίνει μια συνεδρίαση και μια σύντομη ψηφοφορία στο Στρασβούργο. Αλλά αυτό άμα είναι θα γίνει γρήγορα. Αν κατάλαβα καλά λοιπόν, η πρότασή σας είναι να μην προβλέψουμε αυτή την, ε, αυτό το χρονοδιάγραμμα όπως ε, λέει η Γραμματεία, αλλά να περιμένουμε τη συνεδρίαση της Επιτροπής Προϋπολογισμών και των πολιτικών ομάδων, αν κατάλαβα καλά. Ο κύριος ε, Κάλβιν, ε, τι έχει κάνει, έχει πάρει την πρώτα στην καλτιέρη και έχει γράψει το όνομά του πάνω. Εγώ θέλω να γίνουν κάποιες διαγραφές, τα έχω εξηγήσει και στον κύριο Καλτιέρη. Δεν θέλω να καταθέσω τώρα τροπολογίες γιατί άμα ανοίξουμε προθεσμία τροπολογιών θα, θα κινηθεί γρήγορα η διαδικασία. Αλλά εδώ πέρα πρέπει να αλλάξει η πρόταση. Και επειδή δεν το αλλάζει ο κύριος Κάλβιν πρέπει να το κάνουμε εμείς οι ίδιοι. Και, και δεν θα έχει το αποτέλεσμα που θέλουμε η διαδικασία. Πρέπει να έχουμε ένα επικαιροποιημένο έγγραφο, σύμφωνα με την σημερινή κατάσταση των πραγμάτων. Αυτό το πράγμα εδώ πέρα είναι ξεπερασμένο από τα πράγματα. Έχουμε νέα δεδομένα. Εάν δεν το προσαρμόσει αυτό η γραμματεία πρέπει να το κάνουμε εμείς. Ε, δεν θέλω εγώ να κάνω όλη αυτή τη δουλειά. Ε, είμαι και λίγο τεμπέλη, ε, τεμπέλα. Κύριε Πρόεδρε, αν αποφασίσουν οι ομάδες να το ψηφίσουν τον Ιούλιο, θα έρθει η καινούρια πρόταση την ερχόμενη εβδομάδα και θα έχουμε μία ή δύο μέρες προθεσμία για τροπολογίες και θα το ψήσουμε Δευτέρα ή Τρίτη στο Στρασβούργο και θα πάει Τετάρτη στην Ολομέλεια κατευθείαν. Κάλφιν, παρακαλώ. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρέπει εδώ να ακολουθήσουμε την διαδικασία που είναι προς το συμφέρον της Επιτροπής μας. Συμφωνώ με την κυρία Γκρέσλε πως το έγγραφο αυτό ε, δεν λαμβάνει υπόψη τις τελευταίες συμφωνίες. Αλλά πρέπει να προχωρήσουμε ακόμη παραπέρα. Γιατί δεν ξέρω για εσάς, αλλά εγώ δεν είμαι και πλήρως ικανοποιημένο με τα συμφωνηθέντα χτες. Οπότε θα πρέπει να πάμε ίσως και πιο πέρα. Αλλά εάν προτείνουμε να ξαναγράψω εγώ την έκθεση. Εύκολα αυτό γίνεται μέχρι το τέλος της ημέρας. Αυτό σημαίνει πως θα χρειαστούμε και άλλο χρόνο για τις μεταφράσεις. Μετά άλλη μια συνεδρίαση της Επιτροπής, μετά χρόνο για τις τροπολογίες και μετά να συνεδριάσει η Επιτροπή για να υιοθετήσει την τελική έκδοση εκδοχή. Φοβάμαι πως θα πάει η έκθεση στην Ολομέλεια χωρίς τη γνώμη της Επιτροπής μας. Γνωρίζοντα λοιπόν τις ελλείψεις αυτής της γνωμοδότησης, ότι δεν αντικατοπτρίζει τις τελευταίες εξελίξεις, σας, θα κάνουμε αυτά τροπολογίες γιατί αλλιώς η διαδικασία θα πιεστεί πάρα πολύ. Δεν το νομίζω αυτό. Γιατί το ίδιο πρόβλημα είχαμε και με τον κύριο Γκαλτιέρη. και ούτω ή άλλω το ίδιο πράγμα θα μεταφράσουν οι μεταφραστέ για δύο επιτροπέ. Δεν είναι σωστό αυτό το οποίο λέτε. Γιατί το ίδιο πρόβλημα έχει ή Επιτροπή Προπολογισμού. το ίδιο πράγμα θα μεταφράσουν οι μεταφραστέ για δύο επιτροπέ. Δεν είναι σωστό αυτό το οποίο λέτε. Γιατί το ίδιο πρόβλημα έχει η Επιτροπή προπολογισμού. Και λέει, εάν αποφασίσουν την ερχόμενη εβδομάδα κάτι ομάδες θα ψηφιστεί στο Στρασβούργο. Εάν, εάν έρθει. Εάν δεν έρθει ουτω ή αλλω δεν υπάρχει χρονο ε, Οπότε δεν είναι, δεν είναι και αξιοπρεπής αυτή η διαδικασία. Δηλαδή να ασχολούμαστε με ένα παλαιό έγγραφο όταν ξέρουμε πως τα πράγματα έχουν αλλάξει. Εγώ δεν είμαι διατεθειμένη να το επιτρέψω στον εαυτό μου. Το είχα πει και την προηγούμενη φορά. Δεν φταίω εγώ που επελέχθη η διαδικασία που επελέχθη, αλλά δεν μπορώ να δουλέψω, να αλλάξω την παλιά εκδοχή με τροπολογίες. Όχι. Ε, Θα μπορούσαμε να κάνουμε το εξής. Εφόσον η γραμματεία μας κοινοποίησε αυτά που μας κοινοποίησε, ανεπίσημα όμως, όχι επίσημα, θα μπορούσαμε κατά τις προσεχείς ώρες να αποφασίσουμε ότι οι συγητές των σημείων 8, 9 και 10, δηλαδή Κάλφιν, Πάσιτς και Χέρτσοκ, θα έρθουν σε επαφή με την ομάδα εργασίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και με τους συγητές των άλλων επιτροπών για να δούνε αυτό που είπε η κυρία Γκρέσλερ, τι περιθώρια υπάρχουν για να γίνουν οι προσαρμογές ε, σε ε, γρήγορα, ε, όσο γίνεται πιο γρήγορα και τα υπόλοιπα θα μπορούσαν να περάσουν με τροπολογίες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κάνατε μία πρόταση που ήταν ακριβώς αυτό που είχα και εγώ κατά νου. Κάπως αποπροσανατολίστηκα ακούγοντας τον κύριο Κάρπιν και την κυρία Γκρέσλερ. γιατί φαίνεται η κυρία Γκρέσλε, ναι, ε, σαν να ξέρει πράγματα που ο κύριος Κάλφιν, ο εισηγητής, δεν γνωρίζει. Ε, σαν να υπάρχει ε, παραπληροφόρηση. Ε, λοιπόν, εγώ υποστηρίζω την πρότασή σας, Πρόεδρε, να έρθουν όλοι οι υπεύθυνοι σε επαφή μεταξύ τους, να δούμε ακριβώς πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Αυτό δεν αφορά μόνο την Επιτροπή ε, των προπολογισμών και την ε, Επιτροπή Ελέγχου του προπολογισμού. Δεν είναι μόνο αυτές οι επιτροπές που πρέπει να πάρουν μια απόφαση. Καταλαβαίνω την αιτιολόγηση της κυρίας Κρέσλερ που λέει ότι δεν θέλει να κάνει ε, μόνη της όλη αυτή τη δουλειά. Δεν είναι θέμα ολιγορίας. Νομίζω ότι όλοι έχουμε κάποια όρια στην ενέργεια που μπορούμε να διαθέσουμε. Αλλά πιστεύω ότι αυτή είναι μια περίπτωση που δεν θα πρέπει να κάνουμε περιτά πράγματα. Ευχαριστώ. Εντάξει, λέει ο πρόεδρος. Ας προχωρήσουμε. Ας ακούσουμε και τον κύριο Μπάλτσιτης, που είναι ο εισηγητής ε, του σημείου 9, ε, διορθωτικός προϋπολογισμός για την ΕΕ. Παρακαλώ. Ε, Ευχαριστώ. Αγαπητοί συναδελφοί, η κατάστασή μου είναι ίσως πιο εύκολη, εγώ που μιλάω για τον διορθωτικό προπολογισμό, γιατί υπάρχει ένα ποσό, 9 500.000 για το 2010. Το ποσό αυτό έχει μοιραστεί σε δύο κατηγορίες. Είναι 8 εκατομμύρια 870.000 από επιπλέον συνεισφορές των κρατών μελών ε, σύμφωνα με το ΑΕΠ τους και ένα άλλο κομμάτι 645.000 ευρώ υπομορφή φόρων και εισφορών ε, στα συνταξιοδοτικά ταμεία. Η δική μου γνωμοδότηση βεβαίως δεν σχετίζεται με το θέμα που συζητάνε οι κυρίες Γκρέσλε και Κάλβιν. Το είχαμε συζητήσει αυτό και νομίζω πως πρέπει να σημειώσουμε πως ο προϋπολογισμός του 2010 προβλέπει 1625 άτομα παραπάνω προσωπικό από την Κομισιόν και ένα κομμάτι από το Συμβούλιο συν 100 άτομα που θα προσληφθούν. Τα διοικητικά έξοδα θα χρηματοδοτηθούν από την Κομισιόν από 1η Πρώτου του επόμενου έτους. Η υπηρεσία εξωτερικής δράσης θα έχει ένα ξεχωριστό τμήμα όπως συμφωνήσαμε και αυτό θα παραμένει μία από τις βασικές διατάξεις. Αυτές είναι οι βασικές ε, πτυχές ε, που είχαμε συζητήσει Πρέπει να ενισχυθεί ο κοινοβουλευτικός έλεγχος ε, στην εφαρμογή της εξωτερικής ε, δράσης και της ε, ασφαλείας. Πρέπει να χωριστούν επίσης, να διαχωριστούν τα διοικητικά έξοδα, του λογαριασμούς θα τηρεί η Κομισιόν, θα διασφαλίσουμε έλεγχο κοινοβουλευτικό και την διαδικασία της απαλλαγής για τις διοικητικές δαπάνες όπως και για την Κομισιόν και βεβαίως πρέπει να υπάρχει μια ουδετερότητα του προϋπολογισμού να μην υπάρχει δηλαδή αλληλεπικάλυψη της υπηρεσίας αυτής με άλλα θεσμικά όργανα της Ένωσης. Νομίζω πως οι αρχές αυτές ε, θα πρέπει να είναι αποδεκτές και θα δώσω τα έγγραφα προς μετάφραση και μετά θα δούμε ποιες θα είναι οι κατάλληλες προθεσμίες. Ευχαριστώ. Θα μπορούσαμε να περάσουμε στο επόμενο σημείο της δέσμης μέτρων ΕΕΔ, ο κύριος Χέρτσοκ, κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης. Δεν είναι εδώ? Είμαι η κυρία Χέρτσογκ. Αλλά είμαι σε μια κάπως δύσκολη κατάσταση. Εκπροσωπώ την κυρία Χέρτσογκ. Δύσκολη γιατί έλαβα λίγο πριν τη συνεδρίαση το έγγραφο της κυρίας Χέρτσογκ. Γι' αυτό δεν το έχω μάθει ακόμα και έτσι λίγο θα δυσκολευτώ να σας τα πω. Η βάση εδώ πέρα είναι η αλλαγή του κανονισμού που έχει γίνει κυρίως από την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Η κυρία Χέρτσογκ μετά τις πρώτες σκέψεις που αναπτύξαμε στην προηγούμενη συνεδρίαση υπέβαλε σήμερα ένα έγγραφο το οποίο κατ' αναφέρει τα πράγματα τα οποία εμείς θεωρούμε σημαντικά δηλαδή το θέμα, το βασικό θέμα, πώς θα δεσμεύσουμε υπαλλήλου οι οποίοι θα υπηρετούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τι ε, κάτι το οποίο βέβαια είναι πολύ ευκολότερο για υπαλλήλου ε, τη Ευρωπαϊκή Ένωση από ότι για εθνικού υπαλλήλου. Η κυρία Χέρτσογκ προσπάθησε να επεξεργαστεί ε, τα πράγματα τα οποία μπορούμε να κάνουμε εμείς, δηλαδή να υπάρχει μια σαφής αλυσίδα της ευθύνης ε, για να υπάρχει και σαφής ε, ιεραρχία στην απαλλαγή και να δούμε όπως είπα πώς θα είναι και, πώς και η ιεραρχία και η πίστη αν θέλετε στην ε, υπηρεσία και να ξέρουν πώς θα εξοδεύονται και τα χρήματα. Μετά έχουμε ένα νέο εκτιμώντας 4α το οποίο δίνει βάρος στο ότι θα πρέπει να υπάρχει ε, πίστη ανεξαρτησία όλων των υπαλλήλων της ΕΙΕΔ ανεξαρτήτως ε, της προέλευσής τους και κυρίως θα ε, δίνουν λόγο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν θα έχουν ευθύνε έναντι των κρατών μελών που τους αποστέλουν. Και τέλος το θέμα... Α, συγγνώμη, λάθος. Εκτεταμένες διαγραφές που σχετίζονται με το ότι υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία είναι παρεξηγήσιμα όσον αφορά τις ευθύνες, δηλαδή πειθαρχικά ζητήματα και πώς αντιμετωπίζονται, πώς έχει η ιεραρχία... Την, ε, το πώς θα εκδηλώνουν την πίστη τους, αν θέλετε, προς την υπηρεσία υπάλληλη της ΑΕΤ κτλ. Ευχαριστώ κύριε Γκέιερ. Ας περάσουμε τώρα στα σημεία 11, 12 και 13, όπου η συγγετής θα έπρεπε να είναι ο κύριος Ριβελίνη, έχει αντικατασταθεί όμως από την κυρία Γκρέσλερ. Έχουμε το σημείο 11, τροποποίηση του κανονισμού 1605-2002 του Συμβουλίου για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στο Γενικό Προπολογισμό της Ευρωπαϊκής, ε, των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Ευχαριστώ, ζητώ. Συγγνώμη κύριο Ριβελίνη. Ο κανονισμός ο δημοσιονομικός είναι αυτός ο οποίος παρακολουθεί το όλο αυτό κατασκεύασμα και είναι πάρα πολύ σημαντικός για την Επιτροπή μας γιατί πρέπει να ρυθμίσουμε τρία πράγματα. Πρώτα απ' όλα χωρίς αυτόν τον κανονισμό δεν είναι θεσμικό όργανο η ΕΕΔ Οπότε πρέπει να το ρυθμίσουμε κατά τρόπο νόστο στο άρθρο 1, το οποίο υπάρχει και στις τρεις αλλαγές του δημοσιονομικού κανονισμού. Εγώ προτείνω να το κάνουμε μία φορά. Πρέπει λοιπόν να γίνει αυτή η αλλαγή η ίδια παντού λόγω της ε, Λισαβόνας και αναφέρεται βεβαίως ε, μαζί με το Συμβούλιο και η Εξωτερική Υπηρεσία παρά το ότι δεν είναι στα θεσμικά όργανα που αναφέρει η συνθήκη. Οπότε θα γίνει μία φορά αυτή η αλλαγή για να μην το διορθώνουμε συνέχεια και να μην κηρύξουμε τον πόλεμο, αν θέλετε, στο Συμβούλιο. Οπότε αυτό θα γίνει μία φορά. Μετά έχουμε τη σημαντική δουλειά αυτή να ξεκαθαρίσουν οι αρμοδιότητες με την αρχιτεκτονική της υπηρεσίας. Ο πρέσβης ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα διαχειρίζεται τα επιχειρησιακά αυτά κονδύλια σε τρίτες χώρες. Και αυτό είναι πρόβλημα και για εμάς και για το Ευρωπαϊκό ελεγκτικό συνέδριο και το τονίζει αυτό επικριτικά στην έκθεσή του. Οι πρέσβεις λοιπόν αυτοί πρέπει να υποχρεούνται σε κάποια καθάριση ε, λογαριασμών. Οπότε θα πρέπει να δίνουν σε εμά λογαριασμό, λέω εγώ, για το τι κάνουν εκεί πέρα. Η Κομισιόν έχει να κάνει μια δήλωση ετήσια για την διαχείριση των μέσων στις αντιπροσωπείες αυτό είναι κάτι το πολύ σημαντικό το οποίο χρειαζόμαστε και το Συμβούλιο το διέγραψε αυτό, οπότε θα πρέπει να επιμείνουμε όπως και δίποτε. Και θα πρέπει να έχουμε βεβαίω την δυνατότητα να δούμε αυτές τις αιτήσιες δηλώσεις, να βρούμε μια διατύπωση για να έρχονται και σε εμά αν το θέλουμε γιατί υπάρχουν αντιπροσωπείες που διαχειρίζονται πάρα πολλά λεφτά, δίνουν 10% του προϋπολογισμού του αναπτυξιακού. Και ε, να σας υπενθυμίσω τώρα τη συζήτηση που είχαμε για το Αφγανιστάν. Νομίζω καλό είναι να έρχεται ο πρέσβης εδώ πέρα να μας ε, εξηγεί. Κατόπιν διαπιστώνουμε πως υπάρχουν, πρέπει να υπάρχουν γραφές του, του προπολογισμού για την υπατή εκπρόσωπο και οι αποστολές ε, του Συμβουλίου θα πρέπει να δίνουν πολύ πιο λεπτομερή λογαριασμό από ό,τι μέχρι στιγμής. Σκέφτομαι λίγο επίσης, γιατί αυτή η πρέσβη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να δούμε τι δικαιώματα έχουμε αν δεν είναι ικανοποιημένη η Κομισιόν με την λειτουργία. Υπό ποιες συνθήκες απαλλάσσεται από τα καθήκοντά του ο επικεφαλής της ε, αντιπροσωπείας. για να ενισχυθεί αυτή η επιρροή. Καθώς αυτός ο άνθρωπος δεν θα είναι εκεί πλέον στην Κομισιόν, αλλά θα ξοδεύει τα χρήματα της ε, Κομισιόν. Κατόπιν, όσον αφορά την ευθύνη, νομίζω πρέπει να υποχρεώσουμε εδώ πέρα περισσότερο τα κάτι μελη να αναλάβουν την ευθύνη τους. Η ευθύνη είναι πολύ συγκεκριμένη ε, ιστορία Μην ξεχνάμε τον ε, πρέσβη, αν υποθέσουμε, ο οποίος μετά ε, μετατρήθηκε στη Βόρεια Κορέα και δεν μπορούμε να τον αγγίξουμε γιατί έχει και την διπλωματική ασυλία κτλ. Οπότε, οι συνάδελφοι εδώ πέρα θεωρούν πως υπάρχει το δικαίωμα απαλλαγή σε ένα κομμάτι χαρτί και Πράγματι αυτό το έχουμε, αλλά πρακτικά εάν θέλουμε να έχουμε δικαίωμα απαλλαγής, γιατί αυτό δεν υπάρχει, γιατί όπως ξέρετε έχουν μπερδευτεί εδώ πέρα οι αρμοδιότητες. Θα πρέπει λοιπόν να επιμείνουμε, να είναι εφικτό να εξασκήσουμε αυτό το δικαίωμα της απαλλαγής. Κατόπιν, το προσωπικό επίσης ένα πρόβλημα. Τι γίνεται με τους συμβασιούχους πως και αυτοί θα υπαχθούν σε ένα πραγματικό έλεγχο. Κατόπιν διαπίστωσα πως όταν δίνουμε εμείς κάποιο δικαίωμα ελέγχου θα πρέπει να λαμβάνουμε κάτι σε αντάλλαγμα οπότε θα μπορούμε Προσεχώ να προσμετρήσουμε στον προπολογισμό το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης. Μια παλια απέτηση του Κοινοβουλίου που καλό είναι να την έχουμε γραπτός. Και ένα σημαντικό σημείο, ένα από τα λίγα σημεία που δεν με ικανοποιεί με αυτά τα οποία προτείνει ο κ. Γκαλτιέρη, ότι ο εσωτερικό ελεγκτής θα... της Κομισιόν θα είναι και εσωτερικός ελεγκτής της ε, ΑΕΔ γιατί έχει εμπειρία και για να διασφαλιστεί πως η Κομισιόν θα έχει και μια εικόνα του τι γίνεται στην ΕΙΕΔ όσον αφορά την επιχειρησιακή διαχείριση για τον διοικητικό και τον ε, επιχειρησιακό προπολογισμό. Τόσο και κάτι άλλες λεπτομέρειες που είναι ακόμα υποσυζήτηση, αλλά κατά βάση αυτά είναι τα σημαντικά πράγματα. Χρονοδιάγραμμα αυτό και το πότε θα γίνουν οι πληρωμές εξαρτάται από το Συμβούλιο και τον κανονισμό όταν εγκριθεί αυτός ο κανονισμός. Δηλαδή εγώ προγραμματίζω τον Ιούλιο να έχουμε το πρώτο σχέδιο και μετά όταν λάβει απόφαση το Συμβούλιο να ανοίξουμε μια προθεσμία μόλις αποφασίσει ε, το Συμβούλιο. Και να γίνει, τώρα αν θα γίνει πρώτη ή δεύτερη ανάγνωση δεν έχει τόση σημασία. Το σημαντικό είναι στα βασικά αυτά σημεία να έχω την στήριξη των συναδέλφων. Ακόμα κοιτάω τις εφαρμοστικές διατάξεις και το πώς οι πρέσβεις της Ένωσης θα διαμορφωθούν ώστε να γνωρίζουν πως ε, έχουν μια υπεύθυνη ε, θέση. Αυτά και ευχαριστώ. E Ευχαριστώ. Καλύψατε και τα τρία σημεία της ημέρησης διάταξης. 11, 12 και 13, έτσι δεν είναι. Ευχαριστώ. Συγγνώμη. Το σημείο 12. Ναι, 13, όχι, θα συνεχίσω με το 13 ανατριετή αναθεώρηση του δημοσιονομικού κανονισμού. Η αναθεώρηση αυτή υπάρχει εδώ και λίγο καιρό. Είναι το πραγματικά ενδιαφέρον κομμάτι. Και εκεί πέρα θα γίνει πραγματικά η απλοποίηση. Όλα τα υπόλοιπα είναι δευτερεύοντα, ας πούμε. Η Κομισιόν έχει υποβάλει καλές προτάσεις, 180 άρθρα υπάρχουν, 90 ε, επηρεάζονται. Σήμερα το πρωί ε, είχαμε κάποια συζήτηση, είχαμε αυτό το ρίκα στην αναδιατύπωση και σύμφωνα με την συμφωνία του 2009 θα αγγίξουμε μόνο τα άρθρα εκείνα τα οποία έφυξε η ίδια η Κομισιόν. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε εδώ πέρα με την νομική υπηρεσία το εάν πρόκειται πραγματικά περί αναδιατύπωσης και τι χώρο έχουμε για να δούμε και το τι κάνει η Λισαβόνα. Γιατί αν πρόκειται πράγματι περί αναδιατύπωσης, ε, δεν ξέρω αν έχουμε την δυνατότητα να αγγίξουμε όλα τα, τα το πρώτο κομμάτι, το κομμάτι της Λισαβόνα πρέπει να γίνει στο τέλος γιατί είναι αν θέλετε ο όμοιρο τον οποίο χρειαζόμαστε για να έχουμε όντως αυτή την πραγματική απλοποίηση. Γιατί αυτό το οποίο θέλει το Κοινοβούλιο είναι όντως η απλοποίηση. Γι' αυτό σας θέλω πραγματικά να έχετε ε, λίγη υπομονή εδώ πέρα. Δεν μπορώ να κάνω τα απλούστερα πράγματα γιατί θέλουμε να επιτύχουμε κάποιες... Ε, παραχωρήσεις οι οποίες δεν θα γίνουν αλλιώς. Λοιπόν, η τριετής αυτή αναθεώρηση θα είναι μια φιλόδοξη υπόθεση και ο κύριος Ριβελίνη και εγώ ζητήσαμε να υπάρξει μία έκθεση και μία κοινή ε, ψηφοφορία των δύο επιτροπών γιατί ακριβώς προσφέρεται η διαδικασία για να γίνει έτσι, να επιτύχουμε δύο διαφορετικά πράγματα, εφόσον βεβαίως ε, οι αρμοδιότητες είναι στις αρμοδιότητες των επιτροπών μας. Πύχη, να σας δώσω ένα παράδειγμα με το άρθρο 51. Έχουμε το ε, βασικό γνώρισμα αυτής της υπόθεσης η τρίτης. Αυτή η αναθεώρηση νομίζω πως θα πάει στην πρώτη ανάγνωση μέχρι το τέλος του έτους και επειδή αφορά τόσα πολλά άρθρα και επειδή για πρώτη φορά πρέπει να επεξεργαστούμε αυτές τις εφαρμοστικές διατάξεις ταυτόχρονα και είναι δύσκολα τα πράγματα. Οπότε ε, προβλέπεται από την Λισαβόνα κάποια στιγμή την ερχόμενη Άνοιξη να ολοκληρωθεί αυτή η πρόταση γιατί πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα με την Κομισιόν. Υπάρχει μια συμφωνία για τα συγκεκριμένα αποτελέσματα τα οποία βεβαίω και εμείς εδώ πέρα δεν αμφισβητούμε. Οπότε έτσι έχει το χρονοδιάγραμμα αυτή τη στιγμή και νομίζω πως θα καταφέρουμε να έχουμε μια στενή συνεργασία μεταξύ των συναδέλφων Παχόρτ και, και όπως είχαμε και με τον Σλοβαίνο ε, Πρωθυπουργό όταν προσπαθήσαμε να έχουμε καλή συνεργασία. Νομίζω λοιπόν πως με την τριετή αυτή αναθεώρηση έχουμε μια μοναδική ευκαιρία να κάνουμε πιο φιλική προς το χρήστη την όλη διαδικασία. Για να δούμε το τι γίνεται και με τις επιδοτήσεις και με την έρευνα και να ασκήσουμε πίεση στην Κομισιόν έτσι ώστε η αναθεώρηση αυτή να αφορά και τα εξειδικευμένα ταμεία για να δίνει και τον ρυθμό. Γιατί βλέπουμε πως κάθε εξειδικευμένο ταμείο έχει τους δικούς του κανόνες και κάθε απλοποίηση που επιφέρουμε ε, υπονομεύεται από τα ειδικά ταμεία π.χ. τόκι και προχρηματοδότηση εκεί πέρα διαπιστώσαμε πως ε, μπορούμε να μην πληρώσουμε τόκους σε προχρηματοδότηση και ο κανόνας μετά της συγχρηματοδότησης στο Ταμείο Πλαισίου για την έρευνα βλέπουμε πως εκεί πέρα υπάρχουν τόκοι και εκεί γι' αυτό διαμαρτύρονται κατά βάση για την γραφειοκρατία που υπάρχει στην ευρωπαϊκή χρηματοδότηση της ε, έρευνας. Γι' αυτό σημαντικό είναι να δούμε αυτή τη συζήτηση που κρατάει εδώ και χρόνια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 δήλωση εξοπιστίας. Ε, άκουσα τα σχετικά ε, από την κυρία Γκέσλερ. Ξέραμε ε, την ξεκάθαρη πρόθεση της Κομισιόν και της Γενικής Διεύθυνσης ΣΕΤΚΟ που ήθελε να ενισχυθεί ο έλεγχος στους επικεφαλής των αντιπροσωπιών με, σε, σε γενικό βαθμό. Στο Συμβούλιο βέβαια αποδυναμώθηκε λίγο η θέση αυτή διότι καταλήξαμε σε μια διατύπωση που δεν είναι άγνωστη για την ε, βοήθεια, παροχή βοήθειας ε, στο Γενικό Διευθυντή που εκχωρεί αρμοδιότητες. Ωστόσο, η διατύπωση αυτή θεωρούμε ότι είναι αποδυναμωμένη στην προκειμένη περίπτωση. Επομένως, ε, εκτιμούμε την πρόθεση του Κοινοβουλίου να συνταχθεί με τη θέση ενίσχυσης του ελέγχου για το ρόλο που διαδραματίζουν οι επικεφαλείς αντιπροσωπιών. Σε ό,τι αφορά την έκδοση δήλωση αξιοπιστίας. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ευθύνη των προηγούμενων πρεσιών, κάναμε σε βάθος νομική ανάλυση μετά και από τα ερωτήματα που έθεσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι οι κανόνες οι οποίοι θα εφαρμόζονται στους προηγούμενους ε, διπλωμάτες ή προσωρινούς υπαλλήλου. Οι κανόνες αυτοί σε κάθε στιγμή, ακόμη και αν οι υπάλληλοι αυτοί δεν είναι πλέον στην ΕΙΕΔ, θα μπορούν να διώκονται σε περίπτωση που υπάρξει πρόβλημα. Αυτό είναι αδιαμφισβήτητο. Θα μπορούσα ε, διμερώς να μιλήσω με την κυρία Γκρέσλη και να της δώσω τις σχετικές λεπτομέρειες. Σε ό,τι αφορά τον εσωτερικό ελεγκτή, υπάρχει μια διατύπωση που νομίζω ότι κατόπιν πρωτοβουλία του εκπροσώπου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εξευρέθη τελικά συμφωνία. Πρόκειται για μια διατύπωση η οποία κατά την άποψή μας δεν αποκλείει σε ένα άλλο πλαίσιο, όχι απόφασης, θα μπορούσε να συμφωνηθεί ότι ο εσωτερικός ελεγκτής της υπηρεσίας να είναι ο εσωτερικός ελεγκτής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στο σχέδιο απόφασης, το οποίο συζητήθηκε χθε στη Μαδρίτη, κάνει λόγο για συνεργασία. Η συνεργασία βέβαια θα είναι πολύ πιο εύκολη εάν ο εσωτερικός ελεγκτής υπηρεσίας είναι ο εσωτερικός ελεγκτής της Κομισιόν. Αυτό βέβαια δεν αποκλείει τη δυνατότητα ο εσωτερικός ελεγκτής της Κομισιόν να μπορεί να ασκεί αυτά τα καθήκοντα, να παρέχει αυτές τις υπηρεσίες. Ως προς το χρονοδιάγραμμα, το έχω ξαναπεί και εδώ και σε άλλες επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έχω τονίσει ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό οι αποφάσεις να λαμβάνονται γρήγορα. Αν ληφθούν γρήγορε σχετικέ αποφάσεις θα μπορέσει να είναι επιχειρησιακή η υπηρεσία το συντομότερο δυνατό, ήδη δηλαδή από το φθινόπωρο. Είναι ήδη το διάστημα μεγάλο. Σας υπενθυμίζω ότι οι εταίροι μας ε, στις τρίτες χώρες περιμένουν τη δημιουργία της υπηρεσίας αυτής. Εδώ και, χρόνια, και καιρό συγγνώμη, ακούνε να γίνεται λόγος και ανυπομονούν. Δεν πρέπει λοιπόν να καθυστερήσουμε την ε, συγκρότηση αυτής της υπηρεσίας. Χρειάζονται λοιπόν και οι σχετικές νομικές διατάξεις για να μπορέσει να λειτουργήσει αυτή η υπηρεσία. Θα ήθελα τώρα να μιλήσω εν συντομία για την τριετή αναθεώρηση. Χάς, πρόκειται για μια τριετή αναθεώρηση. Και έπειτα, ανατριετία δηλαδή, και έπειτα για αναδιατύπωση, δηλαδή πρώτα τροποποίησης. Είναι σαφές ότι αν επρόκειτο για μία απλή αναδιατύπωση που δεν θα περιλάμβανε ουσιαστικές τροποποιήσεις, τροποποιήσεις της ουσίας του κειμένου, θα ήταν και περιορισμένα τα περιθώρια λιγμών για την κατάθεση τροπολογιών εφόσον επί της ουσίας δεν θα γινόταν τροποποίηση. Στην προκειμένη περίπτωση, επαναλαμβάνω, μιλάμε πρώτα για μια αναθεώρηση. Θεωρούμε λοιπόν σκόπιμο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο πλαίσιο της διαδικασίας να μπορεί να προτείνει τροπολογίες και σε αυτό το χρόνο θα τοποθετείται για αυτές οι Κομισιόν. Σε ό,τι αφορά τώρα τη σχέση μεταξύ του δημοσιονομικού κανονισμού, του γενικού ε, δημοσιονομικού κανονισμού και των τομεακών κανονισμών. Έχω εκφράσει τις απόψεις μου και προηγουμένως και έχω πει ότι εμείς από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποδίδουμε μεγάλη σημασία στην συνέπεια και συνεκτικότητα μεταξύ του Γενικού Δημοσιονομικού Κανονισμού και των τομεακών δημοσιονομικών κανονισμών που θα προταθούν μεταγενέστερα στο πλαίσιο της διαδικασίας για την εκπόνηση του δημοσιονομικού πλαισίου. Όπως είπα και το πρωί στην Επιτροπή Προϋπολογισμών, ο Επίτροπος Αρμόδιος για Προϋπολογισμούς μας έδωσε ξεκάθαρα στοιχεία και ενημέρωσε και τους συναδέλφους του επιτρόπους, δεν υπάρχουν μυστικά. Πολύ ξεκάθαρα λοιπόν τα είπε και ευπέστησε την προσοχή των συναδέλφων του στην ανάγκη να γίνουν σεβαστές οι θεμελιώδεις αρχές που περιλαμβάνονται στο δημοσιονομικό κανονισμό. Και εμείς οργανωνόμαστε κατά τρόπο ώστε ακόμη και χωρίς τη Γενική Διεύθυνση Προπολογισμών, όταν εκπονηθούν οι τομεακοί κανόνες, να συνάδουν αυτοί με τον δημοσιονομικό κανονισμό. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό που είπα θα έπρεπε κανονικά να καθησυχάσει την κυρία Γκρέσλε και όλα τα μέλη της κοινοβουλευτικής αυτής επιτροπής. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Grazie. Ευχαριστώ. Ας περάσουμε τώρα στο άλλο σημείο της ημερήσιας διάταξης σχετικά με τις δυσκολίες των κρατών μελών όσον αφορά τη διαχείριση των διαρθρωτικών ταμείων ε, κατά την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013. Δίνω αμέσως το λόγο στον κύριο Μπλομέιερ ε, που θα μας μιλήσει για την μελέτη που έχει εκπονηθεί και μετά θα δώσω το λόγο στον, ε, στο αρμόδιο μέλος κύριο, κύριο Λιμπεράτσκι. Um, Ευχαριστώ. Θα σας παρουσιάσω πολύ σύντομα μία μελέτη που εκπονήθηκε τους τελευταίους έξι μήνες για διάφορους τομείς της πολιτικής. Τώρα επανερχόμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η μελέτη αυτή αφορά τα διαρθρωτικά ταμεία και πιο συγκεκριμένα τις δυσκολίες των κρατών μελών ε, κατά την ε, οργάνωση των συστημάτων για την περίοδο ε, προγραμματισμού 2007-2013. Πολύ σύντομα, οι τέσσερις τομείς που θα αναφέρω είναι οι στόχοι αυτής της ανάθεσης, η μέθοδος που υιοθετήσαμε, τα ευρήματά μας και κάποια συμπεράσματα, εντέλει και συστάσεις. Καταρχάς, αυτό που μας ζητήθηκε να κάνουμε ήταν να εξετάσουμε τις δυσκολίες των κρατών μελών με ένα κριτικό πνεύμα, αλλά επίσης και ε, προς την κατεύθυνση των λύσεων. Η έμφαση ε, δίνεται λοιπόν στις ε, δυσκολίες που αντιμετώπισαν τα κράτη-μέλη αλλά ταυτόχρονα μας ζητήθηκε να εντοπίσουμε ποιοι είναι οι τομείς εκείνοι όπου μπορεί να υπάρχουν ε, δυνατότητες ε, αλλαγών ε, ώστε να βελτιωθεί η διαχείριση και ο έλεγχος των διορθωτικών ταμείων στο μέλλον. Πολύ σύντομα, ποιο, ποιος ήταν ο λόγος για τον οποίο ανατέθηκε αυτή η μελέτη των δυσκολιών σχετικά με τη διαχείριση και τον έλεγχο. Ένας από τους λόγους και ένας λόγος ανησυχίας που οδήγησε το Κοινοβούλιο ε, στην ανάθεση αυτής της μελέτης είναι η συμμορφώση που γίνεται με πιο αργούς ρυθμούς από ό,τι αναμενόταν ε, για την αναθεώρηση των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου. Η πρόοδος είναι πιο αργή από ό,τι αναμενόταν. Έτσι λοιπόν το Νοέμβριο του 2009 είχαμε περίπου 75% των συστημάτων ε, που είχαν εγκριθεί. Αυτό επηρέαζε και τους ρυθμούς ε, πληρωμών στα κράτη-μέλη και επίσης, αν δούμε στο τέλος του 2009 τα ποσοστά πληρωμών, ε, είναι χαμηλότερα σε σύγκριση με προηγούμενες ε, περιόδους προγραμματισμού. Το 2002, ας πούμε, το συγκρίνουμε με το 2009, βλέπουμε ε, αρκετά μεγάλη διαφορά όσον αφορά την πρόοδο των ποσοστών, των ρυθμών πληρωμής στα διάφορα συστήματα ε, ενισχύσεων. Ε, κάναμε καταρχάς ε, πολύ έρευνα στα δεδομένα που υπήρχαν. Μας διευκόλυνε πάρα πολύ η Κομισιόν παρέχοντας μας πρόσβαση στα στοιχεία αυτά που αφορούσαν τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου των κρατών μελών. Αυτό ήταν ακαδημαϊκή δουλειά. Μετά προχωρήσαμε σε μία έρευνα μεταξύ των ελεγκτικών αρχών των κρατών μελών, 47 ε, ε, ελεκτικές αρχές από 25 κράτη-μέλη συμμετείχαν στην έρευνα αυτή. Επίσης, στη Βουλγαρία, Ισπανία, Γαλλία, Ελλάδα, Λετωνία και Πορτογαλία ε, κάναμε επιτόπιες μελέτες. Αυτό είναι το πράσινο γράφημα που βλέπετε στο κάτω μέρος που δείχνει που είχαμε καλά ποσοστά ανταπόκρισης από τις αρχές. Αυτό ήταν περίπου 50%, ε, 93% των 100 μελών. Και τέλος, ποιες ήταν οι βασικές ερωτήσεις που θέσαμε κατά τη διάρκεια της έρευνας και των συνεντεύξεων που πραγματοποίησαμε. Ποια ήταν η εμπειρία μέχρι τώρα από το κανονιστικό πλαίσιο που θεσπίζει τα συστήματα. Ε, ποια ήταν η εμπειρία σας από την ε, δημιουργία ε, των δομών, των αρχών διαχείρισης, πληρωμής και ελέγχου. Ποιο είναι το ανθρώπινο δυναμικό που χρειάζεται για τη λειτουργία αυτών των συστημάτων. Ποια είναι τα εργαλεία διαχείρισης των πληροφοριών που χρησιμοποιείται. Και τέλος, δύο ακόμα πιο γενικές ερωτήσεις. Πρώτον, θεωρείτε ότι έχει βρεθεί μια ε, ότι έχει βρεθεί ένα σημείο ισορροπίας ανάμεσα στον έλεγχο των διαρθρωτικών ταμείων και την επίτευξη ε, του στόχου ε, της διαρθρωτικής πολιτικής και τέλος ποιες είναι οι συστάσεις για τη μελλοντική περίοδο προγραμματισμού. Αυτό είναι το έγγραφο, το οποίο νομίζω βρίσκεται εδώ στην είσοδο της αίθουσας και αναφέρει λεπτομερώς όλα τα ευρήματά μας και είναι ε, ε, μια απεικόνηση ας πούμε ε, των κυριότερων ευρημάτων μας. Ξεκινώντας από το κανονιστικό πλαίσιο, αυτό που διαπιστώσαμε εδώ είναι ότι για 52% περίπου αυτών που απάντησαν μεταξύ των ελεκτικών αρχών υπάρχουν δυσκολίες, μεγαλύτερες ή μικρότερες δυσκολίες. Για το 15% οι δυσκολίες αυτές ε, ε, είχαν σαν συνέπεια καθυστερήσεις στην εφαρμογή των προγραμμάτων. Ο κυριότερος λόγος ε, των δυσκολιών αυτών, στα πλαίσια δηλαδή του κανονιστικού πλαισίου, ήταν μια αντίληψη ότι οι απαιτήσει δεν είναι αρκετά σαφείς ή ότι υπάρχουν ίσως κάποια κενά και 60% των απαντώντων ε, επισημάναν αυτό το πρόβλημα το πρόβλημα. Όσον αφορά τις ε, ρυθμίσεις για την ε, ε, ίδρυση αρχής διαχείρισης και επιστοποίησης, διαπιστώσαμε ότι ο μόνος τομέας όπου υπήρχε, ε, υπήρχαν θετικές αντιδράσεις ήταν αυτός. Μόνο 35% των απαντώντων ανέφεραν δυσκολίες στον τομέα αυτό, οι οποίες ε, σχετίζονται βασικά με την δημιουργία νέων οργάνων. Είναι ενδιαφέρον να δει κανείς, παραδείγματο χάρη, ότι ε, ο διαχωρισμός ή η σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ των διαφόρων ε, στόχων των διορθωτικών ταμείων δεν φαίνεται να είναι ένα ζήτημα κατά αυτή την ε, περίοδο προγραμματισμού. Ενώ αυτό ήταν ένα θέμα που απασχόλησε περισσότερο κατά την προηγούμενη περίοδο. Τώρα, σχετικά με, τους, με το ανθρώπινο δυναμικό του, τους υπαλλήλους που χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία των συστημάτων και την ποιότητα και την ε, πείρα αυτών των ανθρώπων. Και εδώ έχουμε μια ε, πλειοψηφία των απαντώντων που επισημαίνουν κάποιες ε, ανησυχίες, κάποιες δυσκολίες. Για 40% ήταν μικρές οι δυσκολίες και 18% επισημαίνουν πιο σημαντικές δυσκολίες για την εφαρμογή ε, των πληρωμών. Ένας βασικός παράγοντας που δεν είναι τόσο σημαντικός και δεν προκαλεί μεγάλη έκπληξη ε, είναι ο αριθμός των υπαλλήλων. Ε, γύρω στο 70% των απαντών ανέφεραν ότι ο αριθμός των υπαλλήλων είναι ένα πρόβλημα. Και κατά τις συνεντεύξεις που κάναμε, με φόντο βέβαια την οικονομική κρίση, ε, ε, είδαμε ότι υπάρχουν περιορισμοί όσον αφορά το προσωπικό των ε, δημοσίων διοικήσεων, όμως οι απαιτήσει σχετικά με τους ελέγχους λένε ότι χρειάζεται περισσότερο προσωπικό. Χρειάζεται λοιπόν ιδιαίτερη προσοχή αυτό το σημείο. Τέλος, όσον αφορά τα συστήματα ε, διαχείρισης και επικοινωνίας που χρησιμοποιούνται, εδώ είχαμε το, τις πιο αρνητικές ε, αντιδράσεις. Ε, δύο τρίτα σχεδόν των απαντώντων αναφέρουν δυσκολίες, το ένα τέταρτο αναφέρει σοβαρές δυσκολίες και εδώ είναι οι κυριότεροι λόγοι. Η δημιουργία νέων συστημάτων πληροφοριών. Επίσης, πολλοί κάνουν τη διαφοροποίηση μάλλον πρέπει να επισημάνουμε τη διαφοροποίηση που υπάρχει ανάμεσα στα παλιά και στα νέα κράτη-μέλη όσον αφορά τους περιορισμούς στο προσωπικό που αφορούν ιδιαίτερα τα νέα κράτη-μέλη. Τέλος, όσον αφορά τα συνολικά μας συμπεράσματα, ε, κάναμε τις ερωτήσεις, συζητήσαμε τα θέματα αυτά στις συνεντεύξεις και υπάρχει μια αντίληψη ότι το σημείο ισορροπίας ανάμεσα στον έλεγχο και στο ε, περιεχόμενο δεν βρίσκεται στο σωστό σημείο. Και συνολικά από τις αντιδράσεις που λάβαμε, ε, το συμπέρασμα είναι ότι οι κανονιστικές απαιτήσει κατά αυτή την περίοδο προγραμματισμού ε, έχουν πολύ έντονο προσανατολισμό προς τον έλεγχο και αυτό απομακρύνει την προσοχή από το περιεχόμενο. Κάποια πιο συγκεκριμένα θέματα που προέκυψαν ε, με πολύ έντονο τρόπο είναι παραδείγματο χάρη ότι οι δικαιούχοι αποτρέπονται από τι απαιτήσει του δημοσιονομικού ελέγχου, ότι υπάρχει ε, επιφύλαξη να επιλέξει κανεί ένα project ε, στον τομέα τη καινοτομία λόγω των περιπλοκών που μπορεί να συνεπάγονται οι απαιτήσει ελέγχου και τέλο 70% των απαντώντων έχουν την αίσθηση ότι η διαχείριση των διαρθρωτικών ε, ταμείων αφιερώνει περισσότερο χρόνο στις απαιτήσει συμμόρφωσης ε, και ελέγχου παρά στην επίτευξη ε, των πραγματικών στόχων των προγραμμάτων. Κλείνοντας, ήθελα να πω ότι σχεδόν όλοι οι απαντώντες επισήμαναν ότι θα ήταν απαραίτητο να ε, αντιμετωπιστούν οι δυσκολίες αυτές με περαιτέρω απλούστευση, ούτως ώστε να διευκολυνθεί μια πιο ομαλή διαχείριση και έλεγχος. Ένα άλλο θέμα που φάνηκε πολύ καθαρά είναι ότι είναι σημαντικό σε αυτό το πλαίσιο να μην γίνουν ε, δραματικές αλλαγές, να μην γίνουν θεαματικές αλλαγές ε, και ριζικές αλλαγές, αλλά ε, να γίνουν σταδιακά οι οποιασδήποτε αλλαγές, γιατί χρειάστηκαν πολλές προσπάθειες για να δημιουργηθούν αυτά τα συστήματα. Πρέπει λοιπόν να δοθεί μεγάλη προσοχή στο πώς θα βελτιωθούν αυτά τα συστήματα, ποια θα είναι τα βήματα που πρέπει να γίνουν. Και ένα τελευταίο σημείο από τα συμπεράσματα και από την έρευνα ε, σχετικά με το ποιοι είναι οι τομείς στους οποίους θα πρέπει να ε, δοθεί προσοχή. Ε, πολλές απαντήσεις είπαν ότι θα πρέπει να δίνεται ε, πιο σαφής, πιο έγκαιρη και πιο καθοριστική καθοδήγηση. Η εστίαση πρέπει να γίνεται περισσότερο στο θέμα της απάτης παρά των παρατυπιών. Αυτό είναι κάτι το οποίο προέκυψε σαφώς από τις απαντήσεις. Μετά, σχετικά με τις συστάσεις. η μεγαλύτερη έμφαση καθ' όλη τη διάρκεια αυτών των συζητήσεων ε, δόθηκε στο θέμα της αναλογικότητας. Η αναλογικότητα βεβαίως υπάρχει στον γενικό κανονισμό. Προβλέπονται παραδείγματο χάρη εξαιρέσει ε, για τα πολύ μικρά προγράμματα όσον αφορά τις απαιτήσει που υπάρχουν και αν δούμε τα δεδομένα που έχουμε ε, από τις διαχειριστικές αρχές που διαχειρίζονται μικρά προγράμματα, βλέπουμε ότι ένα πολύ, ένας πολύ μικρός μόνο αριθμός ε, υποφελείται από αυτές τις εξαιρέσεις. Τα ERDF, ε, τα προγράμματα της περιφερειακής ανάπτυξης, έχουν μόνο, από, μόνο 29 από όλα αυτά τα προγράμματα εποφελούνται από αυτές τις εξαιρέσεις. Διότι ε, πολλά από αυτά τα προγράμματα δεν πληρούν ε, το όριο του 40% μέγιστο ποσοστό κοινωτική χρηματοδότησης. Ένας άλλος τομέας όπου έγιναν πολλές συζητήσεις ε, αφορά ε, την, ε, το streamlining ε, σε οριζόντιο επίπεδο του εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου. Αυτό ίσως αφορά περισσότερο τα κράτη-μέλη. Έχουμε την εντύπωση εδώ ότι υπάρχουν πολλές επικαλύψεις. Παρόλο που ο Γενικός Κανονισμός, κανονισμός κάνει σαφώς τη διαφοροποίηση ανάμεσα στις αρχές ε, ε, διαχείρισης, πιστοποίησης και ελέγχου. Πολλές φορές σε εθνικό επίπεδο υπάρχουν επικαλύψεις που σημαίνει ότι επαναλαμβάνονται οι έλεγχοι. Ιδίως αν στα κράτη-μέλη τα διαφορετικά αυτά καθήκοντα βρίσκονται σε διαφορετικά επίπεδα. Παραδείγματο χάρη, ε, υπάρχει μια αρχή ελέγχου σε κεντρικό επίπεδο, ενώ υπάρχουν και τέτοιες αρμοδιότητες και σε περιφερειακό επίπεδο. Και αυτό δημιουργεί ιδιαίτερες περιπλοκές για τα προγράμματα συνεργασία, εδαφικής συνεργασίας, όπου οι διάφορες αρχές ε, έχουν διαφορετικές αρμοδιότητες ε, στα κράτη-μέλη. Ένας άλλος τομέας που αναπτύσσουμε κάπως στην έκθεσή μας είναι το streamlining σε ε, κάθετη κατεύθυνση όλα δείχνουν ότι υπάρχουν ε, πολλές δραστηριότητες ελέγχου που εξετάζουν τα ίδια σημεία των διαφόρων προγραμμάτων. Υπάρχει λοιπόν εδώ περιθώριο περισσότερη, περισσότερη, μεγαλύτερης εξομάλυνσης όλης αυτής της διαδικασίας. Και στις ετήσιες εκθέσεις είδαμε ότι υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αποστολών που πραγματοποιούνται κάθε χρόνο στα κράτη-μέλη. Πέρυσι έγιναν 900 αποστολές ε, πάνω κάτω και οι περισσότερες από αυτές τις ε, αποστολές γίνονται από κοινού με εθνικές ή περιφερειακές ε, αρχές ελέγχου αλλά ε, σε, α, μάλλον είναι, γίνονται σε πολύ μικρό ποσοστό κοινέ αποστολές ελέγχου. Ε, νομίζω ότι η Ολλανδία, ε, η, Τσεχία και η Δανία πρωτοστατούν στην προσπάθεια αυτή κοινών αποστολών ελέγχου. Αλλά όλες αυτές οι αρχές που ερωτήθηκαν θέτουν το ίδιο ερώτημα. Γιατί δεν εντείνεται περισσότερο ε, η προσπάθεια αυτή κοινών αποστολών ελέγχου. Τέλος, πώς θα πρέπει να πραγματοποιηθούν οι βελτιώσεις. Ένα από τα θέματα που ε, επέστησε την προσοχή μας το Κοινοβούλιο είναι ότι ε, υιοθετήθησαν κάποια μέτρα απλούστευσης το 2009 και άλλα πρόκειται να υιοθετηθούν ε, φέτος. Ε, και δεν έχει γίνει συστηματική ε, αξιολόγηση ε, του αντικτύπου ε, των μέτρων αυτών σε κανονιστικό επίπεδο. Ίσως ε, θα πρέπει να ε, ενταθεί περισσότερο η συμμετοχή των κρατών μελών στην όλη αυτή η προσπάθεια. Κάποια στιγμή ζητήσαμε από τις αρχές ελέγχου να μας πούν σχετικά με την εμπειρία τους ε, από τη διαδικασία διαβούλευσης. Ένα τρίτο απάντησαν από τις αρχές ελέγχου ότι έχει ζητηθεί η γνώμη τους. Η πλειοψηφία απάντησε ότι δεν τους έχει ζητηθεί η γνώμη ή ότι δεν βρήκαν το δρόμο τους κατά κάποιο τρόπο μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία απλούστευσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Το λόγο έχει τώρα ο κύριο Λιπεράσχη. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα απλά να πω γιατί ζητήσαμε να γίνει αυτή η έρευνα. Πρώτα απ' όλα υπήρχε το θέμα του ρυθμού απορρόφησης και μετά υπήρχε το θέμα βεβαίω του ποσοστού σφαλμάτων. Και αν δούμε το θέμα του ποσοστού απορρόφησης ε, στο μέσο των δημοσιονομικών προοπτικών ε, του 2003 ήταν γύρω στο 20%, 27%, 30%, 12%. Και είναι ενδιαφέρον αυτό αν δείτε τις δημοσιονομικές προοπτικές ε, και το τι δεν έχει επαναληφθεί σε δημοσιονομικές προοπτικές σε καιρούς ε, κρίσεις ε, βεβαίως που επηρεάζουν τις πολιτικές του προπολογισμού των κρατών μελών και έτσι έχουμε μια εικόνα του τι συμβαίνει καθώς ε, κινόμαστε προς το μέλλον από το 2010 μέχρι το τέλος ε, της περίοδου. Μετά έχουμε το ποστό σφάλματος, αυτό το 12% το οποίο ε, κοιτάμε. Τα καλά νέα νομίζω είναι πως ε, το 2009 είχαμε μια βελτίωση του ποσοστού αυτού και μια αύξηση όσον αφορά την ε, ε, η γενικότερη επιτάχυνση, αλλά το θέμα δεν είναι μόνο το ποστό του φάλματος αλλά και το, η χρήση των κονδυλίων και το να επιτύχουμε τον ε, στόχο μας και είναι ενδιαφέρον να δούμε αυτό το οποίο προτάθηκε αν δούμε δηλαδή τους, ε, το site το ελεγκτικό πρέπει καμιά φορά να δούμε και τις ε, μεθόδους ελέγχου και τα αποτελέσματα. Την ε, ουσία η Κομισιόν εδώ πέρα βεβαίως μας δίνει την δυνατότητα να επιτύχουμε τους στόχους μας μέσω της λογικής χρήσης ε, των κονδυλίων. Αλλά πρέπει να διασφαλίσουμε πως ε, δεν θα χάσουμε και την πλευρά της ε, ουσίας. Θα ήθελα τώρα να περάσω στις συστάσεις ε, που ανέφερε ο πρόσωπος εδώ πέρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Υπάρχουν τέσσερις κατά βάση κλαδί σε οποίους μπορούμε να χωρίσουμε τις συστάσεις και το ποσοστό εκείνο της μη ικανοποίησης που κυμαίνεται γύρω στο 42%. Ε, οι τέσσερις βασικές αυτές τάσεις έχουν πράγματα κοινά, δηλαδή δεν σημαίνει πως είχαμε κάποια επένδυση, αλλά μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και αύξηση του, και ε, του ρυθμιστικού πλαισίου και να είναι σαφείς οι κανόνες, να μην υπάρχει αμφισημία, να βελτιωθεί η επικοινωνία μεταξύ των κρατών μελών και της Κομισιόν και των δικαιούχων. Δηλαδή η συστάση σημαίνει βελτίωση της αποτελεσματικότητας της εργασίας και της πλευράς της οργανωτικής. Τώρα από τη ε, σκοπιά της Επιτροπής Ελέγχου του Προπολογισμού Πρέπει λοιπόν να ξαναδούμε το πώς λειτουργεί όλο το σύστημα και υπάρχει βεβαίως μια πηγή, κάτι το οποίο μπορεί να μας ικανοποιήσει. Βλέπετε πως 64% ε, θεωρούν πως ε, το σύστημα λειτουργεί καλά και δεν χρειάζονται μεγάλες ε, τομές. Πρέπει βέβαια να βελτιωθεί εσωτερικά, να υπάρχει καλύτερη επικοινωνία, περισσότερο προσωπικό και συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και βεβαίως των ε, τελικών χρηστών. Οπότε, με βάση τους στόχους τους οποίους είχαμε θέσεις, θέση, μπορούμε να διαπιστώσουμε πως έχουμε εδώ πέρα μια μελέτη η οποία αφενός απαντάει στο ερώτημα ε, εάν ε, είμαστε αναποτελεσματικοί, αν είμαστε αξιόπιστοι και εγώ θα έλεγα πως πρέπει να δεχτούμε με ικανοποίηση αυτή την έκθεση και να ευχαριστήσουμε τον κύριο Κλωμάγερ και την ομάδα του. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ Γκρέσλε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε κύριε Κλωμάγερ. Πρόκειται για μια καλή μελέτη, αλλά βεβαίως δεν ξέρω τι να πω εδώ πέρα, γιατί τόσοι πολλοί άνθρωποι εφαρμόζουν το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν το καταλαβαίνουν και άρα τι να εφαρμόσουν. Γράφεται πως ε, αξιολόγησαν το ευρωπαϊκό δίκαιο ότι έχει κενά ή ότι δεν είναι αρκετά σαφές. Δοκιμάσατε να τα αντιμετωπίσετε αυτά ή αν έχουν αποκρισταλωθεί κάποιες ομάδες, αν θέλετε, λαθών. Μετά υπάρχει στη σελίδα 32 πίνακας παριθμών 11 και έχω εκεί πέρα ένα ερώτημα. Προφανώς από ό,τι φαίνεται σήμερα ε, έχει μειωθεί ο αριθμός των παρατηρητών, αλλά τα ποσά ε, έχουν αυξηθεί. Οπότε έχουν μειωθεί ο αριθμός των κρουσμάτων, αλλά τα ποσά έχουν αυξηθεί. Μπορείτε να μας πείτε τι γίνεται όχι μόνο με το ΕΤΠΑ αλλά και για τα υπόλοιπα ταμεία. Και τελικά στη Σούμα τι κάνουμε τώρα. Μετά από πέντε χρόνια ε, έλεγχο προπολογισμού, πέντε χρόνια παράπονο για τα διορθωτικά ταμεία, για τα, τους πόρους που δεν ρέουν, τα προβλήματα στην εφαρμογή του ευρωπαϊκού δικαίου. Τι είναι το πράγμα εκείνο που πρέπει να κάνουμε για να ε, βοηθήσουμε λίγο την κατάσταση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Γκάιερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχω κάποια προβληματάκια με την τελική ερμηνεία της ε, μελέτης. Εδώ πέρα συμφωνούμε όλοι πως ε, τα διαρθρωτικά ταμεία πρέπει να οδηγήσουν σε περισσότερη συνοχή ε, στην Ένωση και είναι ένα από τα σημαντικότερα μέσα που έχει η Ένωση στη διάθεσή της γι' αυτό. Διαχειριζόμαστε αυτά τα διαρθρωτικά ταμεία χωριστά. Γνωρίζουμε από τα αποτελέσματα του ελεγκτικού συνεδρίου πως το ποστό σφάλματος είναι πολύ υψηλό και γνωρίζουμε επίσης πόσα σφάλματα κυρίως γίνονται στο επίπεδο των κρατών μελών. Τώρα, κύριε Μπλόμαϊρ, το δικό σας το Ινστιτούτο ρώτησε τα κράτη-μέλη και θα ήθελα να σε να ερμηνεύσετε κάπως τα δεδομένα πιο πολύ από ότι ε, δεν ξέρω από ίσως θα θέλατε, αλλά θέλω να θέσω παρόλα αυτά το ερώτημα. Εγώ δεν ξέρω καμία αρχή που είναι ευχαριστημένη όταν ε, έχει νέους κανόνες. Γιατί κάθε αρχή θα πει ναι, ωραία, τώρα έχω ένα σύστημα. Γιατί καμία αρχή δεν θα πει αχ, τι ωραία. Τώρα θα μου πούνε πω, πω τι σκέφτηκαν πάλι αυτοί οι άνθρωποι. Αυτό θα πει κάθε αρχή. Εξού και αξιολόγηση αυτών των κανόνων με βάση την αποτελεσματικότητά του. Οπότε το ότι το να λένε αυτές οι αρχές πω τι δυσκολεύει η αλλαγή των κανόνων δεν προξενεί έκπληξη. Ε, φυσιολογικό είναι. Ε, κάθε αρχή θεωρεί επιβάρυνση την αλλαγή των κανόνων. Κάθε διοίκηση. Τώρα έχουμε το πρόβλημα πως ε, το υψηλό ποσοστό σφαλμάτων είναι ε, ένας από τους παράγοντες που καθιστούν αναξιόπιστη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί καθόμαστε, ακούμε την έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου στην Ολομέλεια και έρχονται οι ευρωσκεπτικιστέ μας λένε το λάθος ίσον απάτη, άρα μόνο απάτη υπάρχει. Εδώ πέρα δεν λειτουργεί ο μηχανισμός τέλος. Οι μη ευρωσκεπτικιστές βεβαίω εδώ πέρα διαφέρουν. Τα κράτη-μέλη τώρα μα λένε ε, δίνετε τόση βάση στον έλεγχο, συγκεντρωθείτε στην απάτη. Ναι. Αν ε, δούμε τον ρόλο των κρατών μελών, το αντιλαμβάνομαι αυτό, γιατί ε, δεν θέλουν ίσως να υπάρχει τόσος έλεγχος ε, στο τι κάνουν. Και οποιοδήποτε μέλος του ελεκτικού συνεδρίου μετά το δεύτερο ποτήρι κρασί θα μας πει ναι κοίτα τα κράτη-μέλη θεωρούν ότι μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν με αυτά τα λεφτά δικά τους θεωρούν ότι είναι και δεν δίνουν και λογαριασμό και αν είναι να ασχοληθούμε με την καταπολέμηση της απάτης Και διασκεδάζουμε ακόμη περισσότερα γιατί βλέπουμε με πιο ενθουσιασμό και εδώ πέρα βεβαίω ηρωνεύομαι ε, ε, συνεχίζουν τις ε, περιπτώσεις του Όλαφ τα κράτη-μέλη όπου όντως πρόκειται περί καταπολέμησης της απάτης. Δεν το παίρνουν και αυτό πολύ στα σοβαρά. Τελικά έχω την εντύπωση πως ε, εάν θέλουμε να πάρουμε πιο σοβαρά το θέμα της ε, απλοποίησης, νομίζω αυτό θα έπρεπε να χαροποιήσει τις αρχές, εντάξει στην αρχή θα δυσκολευτούν λίγο που αλλάζουν οι κανόνες, αλλά νομίζω η απλοποίηση θα μπορούσε να οδηγήσει στο ότι μειώνεται ο ελεγκτικός φόρτος και αυτό νομίζω θα ικανοποιήσει τους πάντες ε, στο τέλος, αλλά βεβαίω πρέπει να προσέξουμε να μην ξανανεύει το ποσοστό των σφαλμάτων. Για να μην μετατοπιστεί δηλαδή αλλού το, το πρόβλημα. Οπότε το ερώτημά μου είναι εσείς έχετε την εντύπωση στο τέλος αυτής της μελέτης από τα κράτη-μέλη πως ε, ε, θεωρούν τα κράτη-μέλη πως τους ενοχλεί ρε παιδί μου να τους στέλνουν οδηγίες ενέχου από τις Βρυξέλλες. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Τα διαρθρωτικά ταμεία είναι κάτι το πολύ πολύπλοκο, ιδίω για τα νέα κράτη-μέλη, που πριν από μερικά χρόνια ε, άρχισαν να κάνουν πράγματα που δεν τα έκαναν μέχρι τότε και σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Άρα είναι πολύ φυσικό να ε, αντιμετωπίζουν δυσκολίες σε κάποιους ε, τομείς. Υπήρχαν διάφορες ελλείψεις ε, και ελλειπής ενημέρωση, επικάλυψη ε, πληροφοριών. Ε, αυτό όμως ε, είναι του παρελθόντος πλέον. Τώρα περνάμε σε μια νέα εποχή όπου αναλάβαμε το καθήκον να απλουστεύσουμε τα πράγματα. Θα ήθελα να υποστηρίξω λοιπόν τον κύριο Λιπεράσκη που λέει ότι η διαδικασία αυτή θα πρέπει να ευθυγραμμιστεί και να βελτιωθεί και να ε, επιδιώξουμε την απορρόφηση των ε, διαρθρωτικών ταμείων ε, με ένα πιο διαφανή τρόπο. Το πώς θα γίνει αυτό είναι κάτι το αρκετά περίπλοκο. Υπόθηκε ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να συμμετέχουν περισσότερο σε αυτή τη διαδικασία. Πιστεύω όμως ότι θα είναι πολύ δύσκολο τα κράτη-μέλη να απλουστεύσουν τις διαδικασίες για τις οποίες θα είναι υπεύθυνα στο μέλλον. Ε, ίσως θα πρέπει να ακολουθήσουμε ένα διαφορετικό δρόμο. Ε, ίσως θα έπρεπε να δώσουμε μεγαλύτερες αρμοδιότητες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να φέρει εις πέρα σε αυτό το πολύπλοκο ε, καθήκον. Γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γνωρίζει τα προβλήματα που έχουν και τα 27 κράτη-μέλη. Και μόνο αυτή μπορεί να κάνει τις ε, σχετικές προτάσεις πέντε ή 7 κράτη-μέλη ε, να πλουστεύσουν κάποια πράγματα με βάση την εμπειρία των άλλων κρατών μελών. Πιστεύω ότι αυτός ε, είναι ο καλύτερος τρόπος να προχωρήσουμε, ότι θα πρέπει να είναι πολύ ισχυρότερος ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε αυτή τη διαδικασία. Πρόεδρος, έχουμε καθυστερήσει. Δίνω το λόγο για δύο λεπτά για τα συμπεράσματα στον κύριο Μπλο Μέγερ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Αντί για συμπεράσματα θα προσπαθήσω να απαντήσω πολύ σύντομα ε, στους τρεις συναδέλφους που πήραν το λόγο. Η κυρία Γκρέσλε ρώτησε, ε, ζήτησε περαιτέρω πληροφορίες. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες στη μελέτη αυτή. Εγώ προσωπικά ε, εργάζομαι για τη διαχείριση του, των προγραμμάτων του Κοινωνικού Ταμείου και υπάρχουν πολλές ιδέες εκεί, ε, ας πούμε για τα προγράμματα που δημιουργούν εισόδημα. Υπάρχουν πολλές συζητήσεις σχετικά με το πώς θα πρέπει να γίνονται εκεί οι υπολογισμοί. Υπάρχει το θέμα των ε, παραγόντων κόστους. Ε, ίσως υπάρχει μια δυνατότητα εκεί βελτίωσης των ε, κατευθυντήριων γραμμών της καθοδήγησης που δίνεται εξ αρχής. Τα κράτη-μέλη ε, βέβαια δίνουν τις δικές τους ερμηνείες και χρειάστηκε να περάσει αρκετός χρόνος πριν καταλήξουμε σε συγκεκριμένες κατευθυντήρες γραμμές και μια κοινή κατανόηση των διαφόρων ε, ζητημάτων. Όσον αφορά τις παρατυπίες, ε, ίσως αυτό είναι το πιο αδύνατο σημείο της μελέτης μας. Ε, είχαμε την πρόθεση να πούμε κάτι σχετικά με την αποτελεσματικότητα των συστημάτων. Όχι μόνο με τους ρυθμούς πληρωμών και πόσο γρήγορα φτάνουν τα χρήματα στους δικαιούχους, αλλά και ε, σχετικά με τις άλλες πτυχές. Ε, ε στάθηκε εφικτό, παραδείγματο χάρη να περιοριστεί το ποσοστό των λαθών, χάρη στην θέσπιση των νέων συστημάτων. Ίσως έχει, δεν έχει περάσει αρκετός χρόνος ακόμα ώστε να έχουμε τα στοιχεία που να μας επιτρέψουν να συγκρίνουμε ε, τα ποσοστά των παρατυπιών. Τα δεδομένα που έχουμε δεν μας επιτρέπουν να πούμε ότι ναι, ε, το σύστημα δουλεύει, έχουμε ε, μικρότερο αριθμό παρατυπιών ή μεγαλύτερο και να αναλύσουμε τους λόγους. αν λάβουμε υπόψη μας τις σημαντικές καθυστερήσεις που έχουμε την τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού και τα ποσοστά συμμόρφωσης που τα λάβαμε μόλις πρόσφατα, δεν έχουμε αρκετά στοιχεία ακόμα για να κάνουμε αυτή την αποτίμηση. Και κάτι τελευταίο. Δεν προσπαθούμε βέβαια να υποβαθμίσουμε κανένα από τα ζητήματα και από τη διαχείριση των προγραμμάτων ε, που δουλεύω εγώ ε, μπορώ να πω ότι οποιασδήποτε αλλαγέ ενώ μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μπορεί να βελτιώσουν τα πράγματα, ε, πολλές φορές οι άνθρωποι προτιμούν αυτό που ξέρουν από το καινούριο. Αλλά τελικά πιστεύω ότι υπάρχουν ε, ε, πολλοί ε, διαχειριστές των διευθυντικών ταμείων που νοιάζονται για την ποιότητα και για τους στόχους ε, που μπορεί να είναι στους τομείς της καινοτομίας ή της έρευνας ε, και ανάπτυξης. Νοιάζονται πραγματικά και δουλεύουν με συγκεκριμένου περιορισμούς. Υπάρχει ίσως κάποια αντίσταση για, απέναντι στις ριζικές αλλαγές και αυτό ήταν και ε, κάτι που προέκυψε από τις συνεντεύξεις, ε, γιατί δεν μπορέσαμε να κάνουμε σε βάθος ανάλυση ε, στα πλαίσια αυτής της μελέτης, αλλά στις συνεντεύξεις αυτό εκφράστηκε από τις αρχές ελέγχου. Δηλαδή η ικανοποίησή τους ότι δεν ήταν μόνο να ε, απαντήσουν ναι ή όχι και να συμπληρώνουν τα τραγωνάκια, αλλά ότι του ζητήθηκε η γνώμη. Ε, μπόρεσαν να εκφράσουν τη γνώμη τους. Και τα κράτη-μέλη ε, δεν δυσανασχετούν μόνο όταν έρχονται νέοι κανόνες από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και από την εθνική τους νομοθεσία. Και σε εθνικό επίπεδο υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να βελτιωθούν. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος, ε, για αυτά που μας είπατε. Περνάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης, η ειδική έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεκτικού Συνεδρίου ε, σχετικά με την αποτελεσματικότητα της στήριξης του ΕΤΑ για την περιφερειακή οικονομική ολοκλήρωση στην Ανατολική Αφρική και τη Δυτική Αφρική. Δίνω το λόγο στον κύριο Στάς. Ευχαριστώ. Με συγχωρείτε που ήμουν απόν μόνο το απόγευμα, όλη τη μέρα ήμουν στην Επιτροπή Περιβάλλοντος που είχαμε διάφορες ψηφοφορίες και θέσαμε κάποια ερωτήματα και δεν μπόρεσα έτσι να, να φύγω. Η έκθεση αυτή του ελεγκτικού συνεδρίου έχει ήδη συζητηθεί σε άλλη συνεδρίαση και έχει παρουσιαστεί ξανά του Ελληνικό συνεδρίο μου πάλι από αλλά ήμουν άρρωστο και προσπάθησα να κάνω κάπως πιο έντονες ε, τις ε, προτάσεις ε, του ελεγκτικού συνεδρίου. Υπάρχουν εδώ πέρα κάποιες συστάσεις και πρώτα απ' όλα βεβαίως κοιτάμε το τι γίνεται και με το ίδιο το ελεγκτικό συνέδριο και μετά ε, είχαμε και μία συζήτηση και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο διάλογος ε, είχε ως αποτέλεσμα να ξαναγράψω κάποιες από τις συστάσεις μετά από τις απαντήσεις που μου έδωσε η Κομισιόν. Τώρα θα είμαι σαφής, η έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου είναι μία από τις καλύτερες ε, τέτοιες εκθέσεις. Όποιος την διαβάσει ε, εντυπωσιάζεται από το τι γίνεται σε αυτό τον ε, τομέα της ε, πολιτικής. Δεν είναι ικανοποιητική η κατάσταση. Πρέπει πραγματικά να γίνει κάτι. Δεν υπάρχει καθόλου συμπληρωματικότητα μεταξύ εθνικών και περιφερειακών στρατηγικών συνεργασίας της Κομισιόν. Στις συστάσεις μου στο σημείο 2 αναφέρω πως θα έπρεπε η Κομισιόν πριν από τον Οκτώβριο του 2010 να στείλει λεπτομερείς πληροφορίες στη δική μας Επιτροπή εδώ πέρα για τα πράγματα τα οποία δεν πάνε καθόλου καλά και να ζητηθούν μέτρα διορθωτικά για να δούμε λοιπόν το τι θα γίνει το επόμενο έτος αν λάβουμε αυτές τις πληροφορίες τον Οκτώβριο του 2010. Κάτι άλλο το οποίο επίσης προκύπτει σαφώς είναι πως υπάρχει αδυναμία απορρόφησης βεβαίως από την άλλη πλευρά στην Ανατολική και την Δυτική Αφρική και υπάρχει και η ενδιάμεση αξιολόγηση για τις περιφερειακές στρατηγικές στο πρώτο μισό του 2011 και εδώ πέρα απευθύνομαι προς την Κομισιόν πρέπει να λάβει υπόψη αυτά τα οποία αναφέρει το ελεγκτικό συνέδριο και πιθανώς τα ποσά ε, να αναθεωρηθούν. Αυτό μπορεί να είναι προς τα κάτω και προς τα πάνω ίσως, αλλά αυτό θα εξαρτηθεί από την αξιολόγηση. Ανησυχητικό ιδιαίτερα ήταν το ότι σε πάρα πολλές ε, έρευνες ε, το ελεγκτικό συνέδριο δεν μπόρεσε να κρίνει τι έγινε με διάφορα έργα. Όλα αυτά είναι στην ε, σελίδα 40 παράτημα 3 της έκθεσης. Υπάρχει μια σειρά καλών ε, λόγων, αλλά δεν νομίζω πως μπορούμε να το παραβλέψουμε αυτό έτσι εύκολα, καθώς και τη σύσταση πως ε, προ τον Οκτώβριο του 2010 πρέπει να έχουμε κάποια κρίση για αυτά τα έργα που να έχει έρθει στην Επιτροπή μας. Επίσης οργανωτικά θα πρέπει να βελτιωθούν τα πράγματα, να εκπροσωπείται η Κομισιόν σε όλους τους περιφερειακούς αυτούς οργανισμούς και ζητάμε από την Κομισιόν πριν από τον Οκτώβριο του 2010 να μας υποβάλει λεπτομερή έκθεση για το τι έχει κάνει σχετικά με τις συστάσεις του Ελεκτικού Συνεδρίου γιατί συχνά μια καλή έκθεση του Ελεκτικού Συνεδρίου έχει πολύ συγκεκριμένες συστάσεις ε, οι οποίες όμως δεν έχουν μετά καμία συνέχεια και μένουν τα πράγματα μόνο στα χαρτιά, δεν συμβαίνει τίποτα άλλο. Οπότε το ερώτημά μου είναι αν σκοπεύει η Κομισιόν πριν τον Οκτώβριο του 2010 να ε, μας κάνει μια τέτοια έκθεση και ίσως ε, και αυτό πρέπει να το δούμε. Δηλαδή αυτές οι ειδικέ ε, εκθέσεις ε, έρχονται σε εμάς αλλά δεν πάνε στα όργανα του Κοινοβουλίου που ασχολούνται με αυτά τα ζητήματα στην πράξη. Θα έπρεπε π.χ. η ίση κοινοβουλευτική συνέλευση με τις χώρες ΑΚΕ να αφιερώσει λίγη προσοχή σε αυτή την έκθεση και από τις δύο πλευρές, σε αυτή την πλευρά ε, ε, βεβαίως οι ευρωπαϊκοί οι ευρωπαϊκοί εκπρόσωποι, από την άλλη μεριά οι αφρικανοί εκπρόσωποι. Νομίζω πως ε, η διακοινοβουλευτική συνέλευση μπορεί να παίξει ένα θετικό ρόλο εδώ πέρα, ένα ρόλο επικοδομητικού διαλόγου και να φροντίσει πως η περιφερειακή ολοκλήρωση στην Ανατολική και Δυτική Αφρική θα βελτιωθεί, γιατί αυτός πρέπει να είναι νομίζω ένας απόλυτος στόχος για τις χώρες αυτές να συνεργαστούν καλύτερα να επιτύχουν ε, ένα υψηλότερο επίπεδο ολοκλήρωσης. Ένα κομμάτι της Αφρικής νομίζω πηγαίνει καλύτερα από ένα άλλο, αλλά αυτή είναι συνολικά η μεγάλη πρόκληση. Αυτές είναι λοιπόν οι συστάσεις μου και αναμένω παρατηρήσεις ε, και πιθανώς οδηγίες. Βεβαίως εδώ πέρα δεν ψηφίζουμε, αυτό πηγαίνει στον ε, εισηγητή ε, στο τέλος της χρονιάς. Ευχαριστώ. Ο Διευθυντής κ. Κουίν εκ μέρου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ζήτησε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή, τον κύριο Στά, που συναντήθηκε μαζί μα, όπω και αυτό θεωρώ ότι ε, και εγώ ότι ήταν μια πολύ, σύντομη, ε, πολύ χρήσιμη ανταλλαγή απόψεων. Πρώτα απ' όλα πρέπει να πω ότι βλέπουμε την έκθεση και τις συστάσεις του ελεγκτικού συνεδρίου και παίρνουμε τις, την έκθεση και τις συστάσεις ε, πάρα πολύ στα σοβαρά και αρχίσαμε επαφές και με τις δύο αυτές περιοχές. Με την Ανατολική Αφρική πραγματοποιήσαμε σημαντική πρόοδο, ενθαρρύναμε τους περιφερειακούς οργανισμούς να συνεργαστούν περισσότερο και να αυξήσουν το συντονισμό μεταξύ τους. Και πρόσφατα υιοθετήσαμε και μια ομάδα υποστήριξης για να βοηθήσουμε τα πράγματα. Και πράγματι έχει βελτιωθεί η υλοποίηση στην Ανατολική Αφρική. Δυστυχώ η κατάσταση στη Δυτική Αφρική είναι λιγότερο ενθαρρυντική και αυτό είναι ε, ο τομέα και η περιοχή που θα πρέπει να δώσουμε την προτεραιότητά μα στου επόμενου μήνε για να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα τη αποτελεσματικότητα και τη ε, βραδία εφαρμογή. Ερχόμενο τώρα στι συστάσει του εισηγητή, επιβεβαιώνω καταρχά ότι όπω ζητείτε στο σημείο 2, η Επιτροπή τον Οκτώβριο θα δώσει την έκθεσή τη στην Επιτροπή Έλεγχου του Προπολογισμού για το τι μπορεί να γίνει σε ό,τι αφορά τη συμπληρωματικότητα εθνικών περιφερειακών προγραμμάτων, σε ό,τι αφορά τη μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση για του χρόνου, για το σημείο 3. Πράγματι θα δούμε την ικανότητα απορρόφησης και τις επιδόσεις και ενδεχομένω να έχουμε ε, την επιταβελτή επιταχύρω αναθεώρηση. Στο σημείο 4 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Οκτώβριο πάντοτε θα ε, κάνει μια έκθεση για τις ε, περιπτώσεις που δεν μπορέσαμε να αξιολογήσουμε, που δεν μπόρεσε το ελληνικό να αξιολογήσει. Ό,τι αφορά τώρα τους επικεφαλείς των αντιπροσωπιών μπορώ να επιβεβαιώσω ότι τώρα έχουμε αναβαθμίσει την αντιπροσωπεία ε, στο Τζιμπουτί. Είναι πλέον πλήρης αντιπροσωπή. Υπάρχει επικεφάλης αντιπροσωπείας ο οποίος αναλάβει τις σχέσεις ε, με την διακυβερνητική αρχή για την ανάπτυξη, την IGAD. Αυτό σημαίνει ότι όλες οι περιφερειακές οργανώσεις ε, στην Δυτική και την Ανατολική Αφρική έχουν πλέον έναν ειδικό ντόπιο επικεφάλης αντιπροσωπείας. Για το 6 επιβεβαιώνω ότι Αρχές Δεκεμβρίου ε, θα έχουμε μια αναλυτική έκθεση για την Κοκομπού με την συνέχεια που έχουμε δώσει στις συστάσεις μετά την έκθεση του Ενεκτικού Συνεδρίου και ολοκληρώνοντας θέλω να επιβεβαιώσω ότι τις συστάσεις αυτές ε, τις ε, λαμβάνουμε πραγματικά πολύ σοβαρά υπόψη. Σας ευχαριστώ. Grazie. Σας ευχαριστώ πολύ. Αν δεν υπάρχει κάποιος που θέλει το λόγο, νομίζω ότι μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο σημείο Α, παρακαλώ. Ναι, κυρία Γκρέσλε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον ε, κύριο Στάς. Αυτό το οποίο είπε τώρα ο πρόσωπος Κομισιόν είναι, δεν ξέρω, μου εντύπωση καμιά φορά. <sighs> Σκεφτόμαστε το Γαλιλαίο και τον δικό μας ε, μικρό κόσμο, αλλά βλέπουμε εδώ πέρα πόσο μεγάλη είναι η έλλειψη συνεργασίας. Γι' αυτό νομίζω πως αυτό πρέπει να το δούμε και σε σχέση με την υπηρεσία, την ΕΙΕΔ, την υπηρεσία εξωτερικής δράσης ε, και πρέπει εδώ πέρα να μας εγγυηθεί η Κομισιόν που θα παρατηρεί τα πράγματα και θα επιτηρεί τα πράγματα πάρα πολύ στενά. Γιατί, δεν ξέρω, είμαι απεσιόδοξη για την οργάνωση εδώ πέρα. Έχω μία παράκληση πρέπει να ξέρουμε πόσα μέσα εφαρμόζονται, αν θέλετε, από το Αναπτυξιακό Ταμείο στην Αφρική και πόσα από αυτά είναι στήριξη προπολογισμού και ποια είναι διαφορετικά. Θα ήθελα να γνωρίσω λοιπόν ποιοι, ποιους ε, πρέσβεις θα πρέπει εδώ πέρα να στριμώξουμε λίγο αν θέλετε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο εισηγητής για το επόμενο θέμα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω και την κυρία Γκρέσλε που μου επέτρεψε να αναλάβω την εκπόνηση αυτού του σχεδίου έκθεσης. Όπως γνωρίζετε, η έρευνα και η καινοτομία είναι σημαντικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής της Ευρώπης, δηλαδή 2020. Το Συμβούλιο, το ΕΑΡΙΝΟ, υιοθέτησε αυτή την πολύ σημαντική στρατηγική, ένα σχέδιο λοιπόν υπέρ της έρευνας και της καινοτομίας, κυρίως όμως μιλάει για την ένωση της καινοτομίας. Θα έχουμε λοιπόν βελτίωση των διαφόρων ε, συνθήκων πλαισίου για την ε, καινοτομία. Αν θέλουμε να εγγυηθούμε τη μέγιστη δυνατή επίπτωση της πρωτοβουλίας αυτής σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θα πρέπει στόχος ε, να είναι η ελκυστικότητα Θα πρέπει να είναι ανοιχτή δηλαδή η πρωτοβουλία αυτή σε ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, στα πανεπιστήμια και σε όλους τους φορείς της καινοτομία. Αυτό που θα πρέπει να γίνει είναι απλούστευση των προγραμμάτων ανά την Ευρώπη. Υπάρχουν μέτρα απλούστευσης και τα μέτρα αυτά ήδη μας οδήγησαν σε συρρήκνωση των προθεσμιών για τις επιδοτήσεις και για τη μείωση του διοικητικού άχθου για τη διαχείριση των σχεδίων. Σας υπενθυμίζω ωστόσο ότι η δημόσια ακρόασή μα τη 27 η Απριλίου ε, μας είχε οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι η εκπόνηση προγραμμάτων είναι ακόμα περίπλοκη ως διαδικασία. Το παρόν πρόγραμμα πλαίσιο περιλαμβάνει ε, ένα σύνολο μηχανισμών ε, σχετικά με τα ποσοστά επιστροφών, ε, και για διάφορους ε, οργανισμούς. Ο καθορισμός μια σειράς κοινών αρχών στα πλαίσια της διαφοροποιημένης, αντικαθιστώντας τη διαφοροποιημένη προσέγγιση που έχουμε σήμερα, θα οδηγούσε σε σημαντική ελάφρυση των κανόνων, ε, των διαδικασιών και των συστημάτων πληροφοριών. Γι' αυτό ε, είναι αξιέπαινη η ανακοίνωση της Κομισιόν που έχει σαν σκοπό την απλούστευση ε, των προγραμμάτων ε, πλαισίων για την έρευνα. Η ανακοίνωση επισημαίνει τη δυνατότητα περαιτέρω απλούστευσης προς τρεις βασικές κατευθύνσεις. Πρώτα απ' όλα, εξορθολογισμός της διαχείρισης των επιδοτήσεων στα πλαίσια των ισχυών των κανόνων, μέσω βελτιωμένων πρακτικών και διαδικασιών και των μέσων που η Κομισιόν ήδη άρχισε να εφαρμόζει και που θα επιτρέψουν να περιουστεί περαιτέρω ο χρόνος ε, που απαιτείται για τη χορήγηση των υποτροφιών των επιδοτήσεων. Δεύτερον, στα πλαίσια του συστήματος που ισχύει σήμερα με βάση τα στοιχεία κόστους θα μπορούσε να διαθεί περισσότερο, ε, ε, να περισσότερο η μέθοδη υπολογισμού ε, δίνεται στην δυνατότητα επιτάχυσης των διαδικασιών με σκοπό να περιοριστεί ο αριθμός των λαθών που βασίζονται στην προσέγγιση του κόστους. Τρίτον, από την προσέγγιση με βάση το κόστος θα έπρεπε να περάσουμε στην προσέγγιση με βάση τα αποτελέσματα. Κάτι τέτοιο θα μας επέτρεπε να επικεντρώσουμε τους ε, ελέγχους περισσότερο στο τεχνικό και επιστημονικό επίπεδο και όχι στο οικονομικό. Με κατάλληλες ε, διοικητικές ρυθμίσεις ε, για το μέρος της λογιστικής. Υπό το φως όλων αυτών, είμαι ικανοποιημένος με τα μέτρα απλούστευσης και με τις διευκρινήσεις που προτείνονται και επιβεβαιώνω εκ μέρους της Επιτροπής Κοντ την πλήρη υποστήριξη προς τέτοια μέτρα. Σίγουρα, είμαι σίγουρος ότι οι προσπάθειες αυτές θα ε, εξαλείψουν πιθανές ε, ε, διαφορετικές ερμηνείες και προσεγγίσεις και θα αποφύγουμε έτσι την εμφάνιση λαθών. Στα πλαίσια αυτού του νέου προγράμματος πλαισίου θέλουμε ένα σύστημα χρηματοδότησης που ουσιαστικά θα πρέπει να είναι διαφανές, απλό και υγιές. Ένα σύστημα το οποίο θα βασίζεται σε πλήρη εφαρμογή των κανόνων και που θα είναι ικανό να εγγυηθεί την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των ερευνητικών προγραμμάτων στην Ευρώπη. Είναι απαραίτητο να εμποδίσουμε την ε, τροποποίηση των κανόνων κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος, όπως είδαμε κατά το 7ο πρόγραμμα. Διότι θα πρέπει να σεβαστούμε τις ε, νόμιμες προσδοκίες των ε, δικαιούχων. Θα πρέπει να απλουστεύσουμε τον υπολογισμό ε, του κόστους εξαιρώντα το κόστος του προσωπικού για να μην δημιουργείται σύγχυση μεταξύ των συμμετεχόντων. Ε, επιπλέον, και πάντα όσον αφορά το κόστος ε, του προσωπικού που συμμετέχει στι δραστηριότητε έρευνα, το πλαίσιο συμμετοχή σε ένα διαγωνισμό ε, πρέπει τα κριτήρια σχετικά με το κόστος να δημοσιεύονται έγκαιρα ε, ώστε να αποφεύγεται η ασάφεια που πολλές φορές διαπιστώσαμε ότι υπήρχε στα πλαίσια του τρέχοντος 7ου προγράμματος πλαισίου. Τέλος επιμένω ότι στα πλαίσια του, της εκπόνησης του, επόμενου προγράμματος πλαισίου θα πρέπει να έχουμε ένα σύστημα που να βασίζεται στα επιστημονικά αποτελέσματα και όχι μόνο στον λογιστικό υπολογισμό του κόστους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Κάποια σημεία τα οποία θέλω να σχολιάσω για την έκθεση αυτή. Βέβαια βλέπω ότι δεν έχω χρόνο και θα είμαι πάρα πολύ σύντομος. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να επικροτήσω και την έκθεση της Κομισιόν και τη γνωμοδότηση της και να πω ότι αυτό θα αποτελέσει, φαντάζομαι και ελπίζω, ε, τη βάση για τη συζήτησή μας για το 8ο πρόγραμμα πλαίσιο. Πρώτο σημείο που θέλω να σχολιάσω, θα πρέπει πράγματι να υπάρξει εξισορρόπηση μεταξύ του κινδύνου που ενέχεται στην καινοτομία, γιατί δεν συνεπάγεται πάντοτε με την πρόοδο, και την ανάγκη ε, να, σκοπε... να ξοδεύουμε ε, με υπεύθυνο τρόπο τα χρήματά μας. Θα ήθελα να σχολιάσω λίγο την κατάσταση στην Ουαλία όπως λένε οι αρμόδιοι φορείς εκεί, θέλουν να είναι, ξεκάθαροι, να είναι πιο ξεκάθαρα τα μέσα ελέγχου και θα έπρεπε να υπάρχει μεγαλύτερη περίοδος ε, και προθεσμία για, τη, για τους διαγωνισμούς ε, και η εξέβρεση χρηματοδότησης σε, άλλα κράτη-μέλη θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο και μεγάλη βοήθεια. εξέβρεση δηλαδή εταίρων για τη χρηματοδότηση και επίσης η παράταση ε, και του καταπο, της καταποκοπής, το καταποκοπής ποσών και συντελεστών ώστε να μπορούν να αναζητούν, να διεκδικούν το πλήρες κόστος στο μέλλον, αν επεκταθεί η έννοια αυτή. Και τέλος, ε, δύο σύντομα σημεία για τις συστάσεις του εισηγητή. Πρώτα απ' όλα για την παράγραφο 1, όπου καλεί για την απλούστευση, την απλούστευση των μέτρων. Νομίζω ότι θα πρέπει να ορίσουμε επακριβώς τι εστί απλούστευση, τι εννοούμε τον όρο αυτό. Το έχουμε συζητήσει και ξανασυζητήσει στην Επιτροπή μας, αλλά νομίζω ότι χρειάζεται ένας ορισμός της λέξης αυτής. Και τέλος για την παράγραφο 6, όπου ζητείτε ένα σύστημα χρηματοδότησης που θα βασίζεται σε επιστημονικά αποτελέσματα και στις επιδόσεις, στην απόδοση. Νομίζω ότι σκόπιμο θα ήταν να είμαστε λίγο προσεκτικοί. Κατά πόσο αυτό το ερευνητικό έργο θα αποδώσει όχι. Πώς μπορούμε να το κρίνουμε αυτό. Εγώ υποστηρίζω αυτό που λέει παράγραφος, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί για να μην αποθαρρύνουμε καινοτόμα ερευνητικά σχέδια για αυτά τα αποτελέσματα που ενδέχεται να απαιτούνται. Βάζοντα όμω κατά μέρο αυτά τα δύο σχόλια, θα επιβάλλω βέβαια και σχετικά τι τροπολογίε μου, εν γέννη ε, θεωρώ ότι είναι θετική και η γνωμοδότηση και η πρόταση της Ευρωπαϊκή Επιτροπής. Ο κ. Χατζημαρκάκης. Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα να συμφωνήσω με τον συνάδελφο σε αυτό το οποίο είπε. Εγώ είμαι βέβαιο μέλο Ήτρε που ασχολείται κατά κύριο λόγο με αυτή την έκθεση. Και μπορώ να σα πω πω όλα σα τα σχόλια είναι πολύ ευπρόσδεκτα. Αυτό το οποίο πρέπει να λάβουμε υπόψη είναι η ουσιαστική αλλαγή υποδειγμάτων, γιατί μιλάμε για έλεγχο με βάση το κόστος ή πρέπει να περάσουμε σε μια πρόθεση της επιστήμης η οποία θα βασίζεται στην πρόθεση της έρευνας ε, με καταποκοπήν ποσά όπως κάνει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας με πάρα, πολλά καλά, πάρα πολύ καλά αποτελέσματα και με υπέρ αυτής της προσέγγισης. Γι' αυτό θα θέσω εγώ, θα υποβάλω και μια ανάλογη τροπολογία. Επίσης πρέπει να επικεντρωθούμε στην αποτελεσματικότητα της ε, έρευνας πρέπει να θέσουμε στόχους, όχι ενδιάμεσους στόχους, αλλά τους μεγάλους στόχους. Ως ε, στόχους πολιτικής της ε, έρευνας, κάτι το οποίο είναι εξίσου σημαντικό, είναι πως τα ερευνητικά μας προγράμματα δεν είναι ορατά Πρέπει λοιπόν να ασχοληθούμε και με τον έλεγχο γιατί τι γίνεται. Εκεί πέρα διαπιστώνουμε πως όλο και λιγότερο επιστήμονες ζητάνε να χρηματοδοτηθούν από εκεί γιατί είναι πολύ πολύπλοκα. Είχαμε και μια ακρόαση νομίζω σχετική και είναι τρομακτικό το πόσο πολύπλοκα είναι αυτά τα πράγματα τα οποία ζητάμε από τους ερευνητές. Ε, πρέπει να υπάρχει και ένα όριο. γιατί βλέπετε πως μειώνεται η συμμετοχή, ειδικά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Δεν μπορούν να έχουν ένα τμήμα που να ασχολείται μόνο με αυτό. Κάτι το οποίο εγώ δεν βλέπω και θα έπρεπε να υπάρχει είναι ο λεγόμενος ενιαίος έλεγχος, το single audit που λένε. Γιατί υπάρχουν διάφοροι επίτροποι για την έρευνα, δεν είναι μόνο η κυρία Queen, και άλλοι έχουν αρμοδιότητες με άλλες ελεγκτικές διαδικασίες. Δεν είναι δυνατόν, πρέπει να υπάρχει ένας έλεγχος, ενιαίος έλεγχος με αρμόδιο επίτροπο που θα ασχολείται με αυτά τα πράγματα και θα είναι όσο δυνατόν πιο απλός. Αυτό είναι η μόνιμη εποδός. Ευχαριστώ, Γκρέσλε. Σας ευχαριστώ. Ε, πολύ ενδιαφέροντα αυτά τα οποία μόλις είπατε. Θέλω να θέσω ένα ερώτημα. Γιατί δεν υπάρχει κάποια ε, επιτυχία εδώ πέρα, γιατί υπάρχουν ε, πιστοποιητικά μεθόδων τα οποία έχουν εφαρμοστεί. Επίσης θα ήθελα να σας πω πως στην ίδια γενική διεύθυνση δεν είναι δυνατόν διαφορετικοί άνθρωποι να ερμηνεύουν τους ίδιου κανόνες διαφορετικά. Μέσα στην ίδια γενική διεύθυνση. Τουλάχιστον εκεί πέρα πρέπει να βλέπουν τα πράγματα με τον ίδιο τρόπο. Ευχαριστώ. Τον λόγο έχει ο εκπρόσωπος Κομισιόν. Σας ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε τη δυνατότητα να μιλήσω. Θα ήθελα επίσης να εκφράσω τις ευχαριστήσεις μου στην Επιτροπή σας, η οποία μελέτησε αυτό το πολύ σημαντικό αλλά και δύσκολο ζήτημα της απλούστευσης. Συμφωνούμε πλήρως ότι ο πολλαπλασιασμός των χρηματοδοτικών μηχανισμών και εφαρμοστικών ε, οργάνων είναι πηγή πολυπλοκότητας και όλα τα θεσμικά όργανα που συμμετέχουν στην προετοιμασία του επόμενου προγράμματο πλαισίου θα πρέπει να προσέξουν πολύ το θέμα αυτό, να περιορίσουν την πολυπλοκότητα. Θα πρέπει να δουν επίση και την εναρμόνιση ε, των μεθόδων εφαρμογή μεταξύ των διαφόρων εργαλείων και οργανισμών και μηχανισμών. Σε ό,τι αφορά τώρα τη συζήτηση για την προσέγγιση βάση αποτελεσμάτων και την πιο εντατική χρήση των καταποκοπήν ποσών, ε, είμαστε ευγνώμονε για το ότι η Επιτροπή σα φαίνεται να καλωσορίζει την προσπάθεια αυτή τη απλούστευση. Ωστόσο, θα πρέπει ταυτόχρονα να επιστήσω την προσοχή σας στο ότι υπήρξαν κάποιες αντιδράσεις που λάβαμε για την πρόταση από πολλούς ενδιαφερομένους φορεί αλλά και από ευρωπαϊκού ευρωπαϊκούς φορείς, ευρωπαϊκά, ευρωπαϊκούς οργανισμούς και φαίνεται να μην πρόκειται πια και για την πανάκια ε, σε καθολικό επίπεδο. Εξεφράστησαν δηλαδή ανησυχίες και ακούσαμε και από εδώ ε, κάποιες ανησυχίες. Ίσως λοιπόν γίνει σταδιακή εισαγωγή για να δοκιμάσουμε τις προσεγγίσεις ε, αυτές με πιλωτικά προγράμματα και μετά να προχωρήσουμε σε γενικότερη εφαρμογή. Σε ό,τι αφορά τώρα τα συγκεκριμένα ερωτήματα σε σχέση με τα πιστοτικά για τη μεθοδολογία. Νομίζω ότι εδώ θα πρέπει να κάνουμε τη διάκριση μεταξύ δύο περιπτώσεων. Το πρώτο είναι το προσωπικό για το μέσο κόστος προσωπικού και το δεύτερο είναι το πιστοποιητικό του χρήστη. Σε ό,τι αφορά τη δεύτερη περίπτωση, για τα όργανα που δεν χρησιμοποιούν το προσωπικό, για το, μέσο κόστος, το πιστοποιητικό για το μέσο κόστος προσωπικό, είναι σχετικά μικρός ο αριθμός των πιστοποιητικών που εγκρίνονται. Ένας λόγος μπορεί να είναι ότι η προστιθέμενη αξία για το είδος αυτό του πιστοποιητικού δεν είναι πολύ μεγάλη. Το... Πρόκειται για κάποιο μέρος του κόστους του ενδιάμεσου προσωπικού. Σε ό,τι αφορά όμω την άλλη μεθοδολογία για το μέσο κόστο προσωπικού, εκεί το ζήτημα είναι πιο πολύπλοκο. Συγκεκριμένα σχετίζεται με το συνολικό ε, πλαίσιο λογοδοσίας. Έχουμε το... την ετήσια δήλωση εξοπιστίας, έχουμε ε, τα διάφορα ετήσια όρια και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ορίσει τα κριτήρια επιλεξιμότητας ε, για την μέθοδο αυτή του μέσου κόστους, ακολουθώντας τη γενική προσέγγιση. Στην ανακοίνωσή μας για την απλούστευση έχουμε προτείνει μια πιθανή διέξοδο γιατί γνωρίζουμε ότι η κατάσταση αυτή δεν είναι δυνατό να συνεχιστεί έτσι. Σε έναν βαθμό η προτινόμενη αλλαγή θα απαιτήσει αλλαγή των κανόνων συμμετοχής, αλλαγή δηλαδή του νομοθετικού πλαισίου, του 7ου προγράμματος πλαισίου. Θα μπορούσαμε να εξετάσουμε το ενδεχόμενο ε, να επιλύσουμε αυτό το πρόβλημα αλλάζοντας ολόκληρη την προσέγγιση και από αυτήν την έννοια θα είμαστε γνώμονες στο Κοινοβούλιο και στην Επιτροπή σας συγκεκριμένα αν εγκρίνατε ρητός την αλλαγή αυτή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής θα γίνει στις 12 Ιουλίου στις 3 η ώρα. Τώρα, ε, για κλεισμένο το θηρόν, θα γίνει η συνεδρίαση των συντονιστών. Ευχαριστώ.